Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Let me open our... Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Επιτρέψτε μου να κηρύξω την έναξη συνεδρίασής μας. Ο πρόεδρος κύριος Μπροκ είναι καθοδόν. Τον καθυστέρησαν κάποιες σημαντικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει. Effectively, I will be... Και για να αξιοποιήσουμε το χρόνο θα προεδρεύσω προσωρινά βέβαια και θα αναλάβει μόλις καταφτάσει, ελπίζω να μην το πειράζει. Σας ευχαριστώ. Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση του σχεδίου τη ημερήσια διάταξη. Πρέπει να σα ενημερώσω ότι έχουμε δύο αλλαγέ. Ο Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν ματέωσε τελευταία στιγμή την επίσκεψή του στην Ευρώπη και πρέπει να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη. Ανταυτού λοιπόν, που είναι το σημείο 7, έχουμε τώρα ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες που έγιναν για το ψήφισμα της Σερβίας. Το αρχικό θέμα 9, όπως είχε προγραμματιστεί. Κύριο κύριος Τάνο, εισηγητής μας για το Μαυροβούνιο, ασθενή. Το θέμα του θα το συζητήσουμε λοιπόν το απόγευμα. Αφού σας τα είπα αυτά, αρχίζουμε τη συνεδρίαση. με το θέμα υπάρχουν τέσσερα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση πρόοδου για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη 2011. Ε, η συγκήτριά μας είναι η κυρία Πακ και της δίνω μέσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που αντικαθιστάτε τον κύριο Μπροκ για να αρχίσουμε γρήγορα γιατί πρέπει να πάω να ψηφίσω σε άλλη επιτροπή. Σας παρακαλώ να με συμπαθάτε λοιπόν. Δεν θα επαναλάβω όλα αυτά που είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση αλλά θα επικεντρωθώ σε αυτό που καταφέραμε χτες να συμφωνήσουμε ε, ως συμβιβασμό με τις συναδέλφους, γιατί μόνο κυρίες ε, ήταν. Από τότε που κατέθεσα εγώ την πρότασή μου έχουμε θετικές εξελίξεις στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν επιτρέπεται να ονομάζεται κυβέρνηση αλλά Υπουργικό Συμβούλιο. Για μένα το ίδιο είναι, τουλάχιστον αυτό ελπίζω και συμφώνησαν να ρυθμίσουν ε, τα θέματα που εκκρεμούν ακόμα. Έχει ήδη εγκριθεί ο νόμος περί απογραφής. Δύο πράγματα εκκρεμούν από τα πέντε συν δύο σημεία που πρέπει να διεκπαιρεθούν ακόμα, όπως είπε ο υπέτος εκπρόσωπος. Και αυτό είναι το ένα η ιδιοκτησία του στρατού και η κρατική ιδιοκτησία. Αυτά τα δύο πρέπει ακόμα να λυθούν. Και από εκεί και πέρα είναι έτοιμη η Βοσνία Ζεγοβίνη να μπει στο δρόμο προς την Ευρώπη και το σύμφωνο σταθεροποίησης και ε, συνεργασίας και σύνδεσης και περί τα τέλη του χρόνου να κάνει ε, και αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι είπε ο επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου. Βέβαια μέχρι τότε θα περάσει πολύ καιρό και θα κυλήσει πολύ νερό στο ποτάμι, όπως πάντα κυλούν τα ποτάμια στα Βαλκάνια. Ε, πάντως έχουν δηλώσει προθυμία να δημιουργήσουν τους θεσμούς και τα προβλήματα που έχουν να λυθούν να μπω λίγο στα επίμαχα σημεία, θέλετε, που υπήρξαν στην έκθεση, τα οποία όμως στο μεταξύ ελπίζω να έχουν ε, λυθεί και αποσοφηθεί με διατύπωση που να συμφωνούν όλοι για να την δέχονται. Το πρώτο. Τι να γράψουμε ότι ο ύπατος εκπρόσωπος θα πρέπει τώρα να αποχωρήσει από τη χώρα. Εγώ το έβαλα πάρα πολύ ε, προσεκτικά στην έκθεση, να το κοιτάξουμε, να το μελετήσουμε, να το εξετάσουμε. Πολλοί συνάδελφοι όμως θέλησαν να πούν ότι υπάρχουν προϋποθέσεις. Θυμίζω αυτές τις πέντε συν δύο. Δυστυχώς πριν από χρόνια είχε δοθεί αυτή η δέσμευση και η υποχρέωση και ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Βρήκαμε τελικά μια διατύπωση όμως ε, που να ανταποκρίνεται και στην επιθυμία μας να αποχωρήσει από τους εκπρόσωπους γιατί δεν είναι ε, πλέον απαραίτητο. Θα πρέπει να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους οι άνθρωποι εκεί, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθούν αυτά τα σημαντικά που πρέπει να υλοποιηθούν. Ε, και στην πρότασή μου λέγω θυμίζει ότι οι αρχές Βοσνίας ζεγοβίνης θα πρέπει σε αυτά τα πλαίσια να λύσουν τα εκρεμή ζητήματα που αφορούν την ιδιοκτησία του κράτους και των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή οφείλουν. Είναι προϋποθέσεις, αλλά είναι καλό να μην αναφέρεται η λέξη προϋποθέσεις. Συμφώνησαν οι συνάδελφοι χτες λοιπόν να προχωρήσουμε έτσι. Τώρα, έχουμε ένα άλλο μικρό πρόβλημα στην προστασία των μειονοτήτων. Είχα μια λάθος διατύπωση, εγώ φταίω γι' αυτό. Τώρα έχουμε εντάξει ομάδες και άτομα, ε, groups και individuals και με μονομένα πρόσωπα. Άλλο θέμα που χρειάστηκε συμβιβασμό και είχαμε πρόβλημα. Την περασμένη φορά δεν κυριάρχησε, αλλά ο κύριος Μπέλτερ ε, ανέφερε το θέμα των ε, Ουαχαβητών και αυτό οδήγησε σε μεγάλη φασαρία ε, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και βγήκε η Ρεπούμπλικα Σέρψκα και ο τύπος εκεί και μου, ε, απέδωσε διάφορες δηλώσεις ότι είχα πει εγώ λέω ο μεγάλος μουφτής εκεί ήταν ε, εκπρόσωπος αυτών των Ισλαμιστών και τα λοιπά και είχαν παρακολουθήσει όμως τη συνεδρίασή μας και στο διαδίκτυο και μπορούμε να τους παραπέμψουμε σε αυτή. Τελικά στο Σαράγεφο υπήρξαν όμως ε, και ε, δημοσιεύματα ότι εμένα με πληρώνει με δοτή του κυρίου Ντόντικ, ο οποίος ο κύριος Ντόντικ ανέκαθεν με καθίβρισε. Καταλαβαίνετε τα πράγματα και πώς ε, τα αντιλαμβάνονται εκεί. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως αυτό το θέμα των Ουαχαβίτ ε, παραμένει γιατί οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη και μέσω της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Είναι μια οργάνωση εντός του Ισλάμ πάρα πολύ ακραίων στοιχείων, τους οποίους φοβούνται και στον αραβικό κόσμο. Όχι όλοι, είναι μια ομάδα, πώς να το πω, ένα ρεύμα του Ισλάμ που έχει φύγει από τη Σαουδική Αραβία και φτάνει και στο ε, ε, Ιράν και στο Ιράκ και εκεί το, το φοβούνται αυτό το κίνημα και τελικά εγώ δεν θέλω στη Βοσνία και τελικά στο Κόσοβο αργότερα γιατί έχουμε το ίδιο πρόβλημα να ε, εκπληρώσει αυτό που έλεγε ο Μιλόσεβιτς στην αρχή ε, αυτών των αγριοτήτων που έκανε ότι θέλει το Ισλάμ να μας κυριεύσει και μας απειλεί εάν στα Βαλκάνια, στο Κόσοβο, στη Βοσνία ή και στη Σερβία ε, εδρεωθούν οι Γουαχαβίτες, είναι μεγάλη απειλή. Θέλω να σας διαβάσω όμως ακριβώς την παράγραφο πώς το έχουμε διατυπώσει για να μην θεωρεί κανείς ότι ε, επιτιθέμεθα σε οποιουσδήποτε μουφτίδες ή ε, ε μουσουλμάνους. Και πριν έρθει το τσουνάμι θα πρέπει να το σταματήσουμε. Έλεγα λοιπόν ε, στο συμβασμό 8, καλεί τις αρχές της Βοσνίας να καταπολεμήσουν τον εξτρεμισμό, τη μυσαλλοδοξία και τη βία σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Ανησυχεί για ε, τις ακραίες εκφάνσεις των ΟΑΧΑΒΙΤΟΝ και όπως και άλλες ε, ακραίες τάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Καλωσορίζει την το κήρυγμα της Παρασκευής του Μεγάλου Μουφτή του Νοεμβρίου του 2011 που ε, καταδίκασε την τρομοκρατία και τη βία ως ε, εχθρικές πράξεις, ε, πράξεις συγγνώμη, κατά του Ισλάμ και τα λοιπά. Καλή τη διερεύνηση, την επαγρύπνηση και την απομάκρυση κάθε είδους εξτρεμιστικών απειλών στην περιοχή. Νομίζω ότι το δέχονται οι συνάδελφοι, είναι ο συμβασμός υπαριθμών 8. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι κατά αυτής της διατύπωσης. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι προσπαθούμε ε, να πούμε προσοχή. Έχω και μια προφορική τροπολογία. Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί οι πολίτες ε, του Κωσυφοπεδίου και οι Βόσνοι που ζουν στο Κωσυφοπεδίο εδώ και τρία χρόνια πια δεν μπορούν να πούν στη Βοσνία από πουθενά. Κανείς δεν αναγνωρίζει την ταυτότητά τους ούτε το διαβατήριό τους. Είναι η μόνη χώρα. Ακόμα και η Σερβία. Ακόμα και η Σερβία δέχεται τις ταυτότητες του Κωσυφοπεδίου. Και όλες οι χώρες ακόμα και εκείνες που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο ε, κράτος, ε, δέχονται όμως την ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο ή το διαβατήριο. Εκτός από τη Βοσνία, είναι η μοναδική χώρα που δεν το επιτρέπει. Ε, παρακαλώ συμφωνήστε να κάνουμε ε, προφορική τροπολογία, ε, μια στιγμή να τη βρω, ανησυχεί που η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι η μόνη χώρα της περιοχής που δεν επιτρέπει την είσοδο πολιτών του κοσυφοπεδίου στην επικράτειά της. Καλεί λοιπόν τις αρχές της χώρας να εγκρίνουν τα απαραίτητα αυτά ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως ο πράττουν άλλωστε η Σερβία και άλλες χώρες της περιοχής. Ελπίζω να συμφωνείτε. Και ένα δεύτερο μικρό πρόβλημα έχω ακόμα. Και αφορά τις τροπολογίες κυρίας Μποσκούρτ για τα θέματα των συνόρων. Γνωρίζετε ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει ε, μεγάλα μακριά σύνορα με τους πάντες περίπου στην περιοχή. Και εγώ δεν ήθελα την τροπολογία της κυρίας Μποσκούρτ που είναι μεγάλη και μακροσκελής, δεν ξέρω αν συμφωνεί, αλλά προτείνω το εξής. Εμείς δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε στη Βοσνία με ποιο τρόπο θα λύσει τις μεθοριακές διαφορές με τους γείτονές της. Με διατησία, με συνθήκη, έχουν δοκιμάσει τα πάντα μέχρι τώρα στην περιοχή, αλλά ναι, εκτό από πόλεμο ακόμα. Και είπαμε καλεί την κυβέρνηση Βοσνίας Ερζεγοβίνη και τι γειτονικέ χώρες να κάνουν ό,τι μπορούν για να λυθούν οι ε, μεθοριακέ ε, διαφορές. Με την Κροατία το κάναμε. Δεν χρειάζεται να την κατονομάσουμε. Αφορά τη Βοσνία και τους γείτονές της. Και θα πρέπει για την έκθεση για την Κροατία, να το αναφέρουμε αυτό στην έκθεση αυτή σε ό,τι αφορά την Κροατία. Αυτά ήταν τα πιο προβληματικά σημεία. Ναι. Και κάτι άλλο που προσθέσαμε μετά την τροπολογία της κυρίας Κορνέλησεν και το κοινό στα γερμανικά πάλι το γραφείο του υπάτου εκπροσώπου του κυρίου Σόρενσεν που είναι ο πρέσβης μας βασικά εκεί είναι και καλός, προσφέρεται για την περιοχή. Ε, θα πρέπει να ενισχυθεί το γραφείο του στην περιφέρεια. Δεν αρκεί μόνο να είναι η παρουσία του στο Σαράγεβο. Στην Πανιαλούκα, Λούκα, στο βορρά, έχουμε ένα γραφείο, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή στελέχωση. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει έναν οδηγό μόνο. Είπαμε ότι θα πρέπει να επεκταθεί και να αυξηθεί το προσωπικό και στην Πανιαλούκα να είναι περισσότεροι και στο Μόσταρ αλλά εχθές στη συζήτηση με τον κύριο Σόρεσεν ακούσαμε ότι πρέπει να πάμε και στην Τούσλα γιατί ε, είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας γιατί εκεί υπήρξε ένας δήμαρχος τον Πέσλαγκης, τον θυμάται ε, κανείς από εσά. Ε, και σε δύσκολους καιρούς ήταν πάρα πολύ εξαιρετική η δράση του και η παρουσία του. Θέλουμε λοιπόν ο, ο εκεί, ο, εκπρόσωπός μας να έχει και περισσότερο προσωπικό και μεγαλύτερη στελέχωση. Και αν φύγει ο διεθνή τους εκπρόσωπο, μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε και προσωπικό να βρούμε εκεί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ του συντονιστέ για την τόσο καλή συνεργασία και σας παρακαλώ να μην το συζητήσουμε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να πάω στην Επιτροπή Πολιτισμού να ψηφίσω. Ευχαριστώ. Κυρία Πακ, σας ευχαριστώ πολύ που μας αφιερώνετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα καταβληκτικά σας αγγλικά που ακούσαμε μόλις τώρα. Μάλιστα. Ήμουν στο Ιρλανδικό μέτωπο σήμερα το πρωί Έδωσα συνέντευξη στο Ιρλανδικό ραδιόφωνο ε, για το θέμα του δημοψηφίσματος. Όπου δεν έχουμε δυσκολίες πάμε και τις ε, βρίσκουμε μόνοι μας. Η κυρία Μποσκούρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι καλό που έχει προκύψει τώρα νέα κυβέρνηση, ακόμα και δεν την λένε κυβέρνηση, ε, που θα επιταχύνει όλα αυτά τα ζητήματα και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Καλό που εγκρίθηκε ο νόμος για τις κρατικές ενισχύσεις και για ε, την ε, απογραφή, αλλά θα πρέπει να υλοποιήσει και τις 7 δεσμεύσεις από τη Συμφωνία του Dayton, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους εσωτερικούς πρόσφυγες και εκτοπισμένους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που χρειάζονται ε, για να προσαρμοστεί η νομοθεσία με τις αποφάσεις του δικαστηρίου και να γίνει ένα λειτουργούν κράτος. Η Βοσνία Ερζεκοβίνη μπορεί να μπει στην Ένωση μόνο σε ενιαία χώρα, θυμίζω. Για τους Ουαχαβίτες έχουμε συζητήσει πολύ. Δυστυχώς αυτό το θέμα είναι κρίμα από κυριαρχή στον τύπο, γιατί οι Ισλαμικές κοινότητες στη Βοσνία Ερζεγοβίνη το θεωρούν εξίσου ανισχυτικό και θέλουν να πάρουν τις αποστάσεις τους από όλους αυτούς. Ε, δηλαδή, δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή την ομάδα και να δυσμονούμε ότι υπάρχουν και άλλες εξτρεμιστικές τάσεις παντού ε, στα Βαλκάνια ε, εθνικιστών. Οι συμβιβαστικές τάσεις τώρα είναι ε, ε, εντάξει και μπορούμε να τις υποστηρίξουμε, ελπίζω. Για την Κροατία, πραγματικά, είναι πολύ μεγάλα τα σύνορα και ε, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν, είναι σημαντικό. Γι' αυτό έχω κάνει τη δική μου τροπολογία. Θα την ψηφίσουμε χωριστά. Ελπίζω να μπορέσετε να την υποστηρίξετε. Είναι σημαντικό η Ελλάδα και η είναι ε, σημαντικό συγγνώμη, η Κροατία και η ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη να τα βρουν ως καλοί γείτονε. Και όταν γίνεται λόγος για συμφιλίωση θα πρέπει τα θύματα βιασμού κατά τη διάρκεια του ε, πολέμου να δικαιωθούν και να συμμετέχουν όλα τα μέρη σε μια στρατηγική στη τροπολογία μου έχει ζητηθεί τη ψηφοφορία. Ελπίζω τα περισσότερα τμήματα να μπορέσει και η συγγήτρια να τα δεχτεί. Χθε ο κύριος Σόρενσεν επιβεβαίωσε ότι ε, χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή και βοήθεια ε, από εμά και τα θύματα. Αλλιώς δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ορισμένα ταινίε δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ την κινηματογραφική ταινία της κυρίας Αντζελίνα Τζολί. Επίσης, να αλλάξει ο νόμος για την ηθαγένεια, όπως ζήτησε ε, το συνταγματικό δικαστήριο. Είναι επίγον αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατσίν έχει το λόγο. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω σλοβενικά, τη γλώσσα μου. Ευχαριστώ. Η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι μια χώρα περίπλοκη και πάρα πολύ ευαίσθητη. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ισορροπημένοι και πάρα πολύ προσεκτικοί στις δηλώσεις μας. Ε, έγινε λόγος για τους Βαχαμπίτες και μετά έγινε χαμός με μικρή αφορμή και ασχολούμαστε σε αυτή τη συζήτηση με αυτό το φαινόμενο που είναι πάρα πολύ περιορισμένο και το περιστατικό και το επεισόδιο που έγινε πριν από λίγο καιρό εντάξει, εντοπίστηκε κάποιος ένοπλος, αλλά η Βοσνία ε, Ερζεγοβίνη είναι η δημοκρατία των Δυτικών Βαλκανίων με ε, σαφή δημοκρατική προοπτική. Δεν είναι Σαουδική Αραβία. Η 8η ε, συμβιβαστική τροπολογία είναι κατά τη γνώμη της ομάδας μας ισορροπημένη και μπορούμε να τη δεχθούμε. Υπάρχει μια τροπολογία που ζητεί μια ειδική διάσκεψη η Βοσνία Ζεγοβίνη πρέπει να κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό της ε, για τη συμφιλίωση. Το θέμα δεν είναι μόνο η απόφαση Σέντιτς Φίνση για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να εκπροσωπούνται στην Προεδρία. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Θα πρέπει να είναι μια χώρα και ένα κράτος που να μπορεί να λειτουργεί. Ε, ορισμένοι θεωρούν ότι ε, θα πρέπει να φύγει ο ύπατος εκπρόσωπος. Εγώ είμαι λίγο πιο επιφυλακτικός εδώ. Νομίζω η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να διατρανώνει περισσότερο τη φωνή της του εκπροσώπου της εκεί. Όταν κάποιος ανείται τη Γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα, τι γίνεται. Ε, εδώ συζητούμε για τους Γουαχαμπίτες, αλλά δεν έχουμε συζητήσει το θέμα της Σρεμπρένιτσα. Δεν ε, ε, έχουμε ένα τρόπο να τιμωρούμε εκείνους που αρνούνται αυτή τη γενοκτονία και αυτό θα κάνει αδύνατη τη συμφιλίωση. Και εγώ υποστηρίζω ε, τις προσπάθειες του κυρίου Σόρεσεν να ενισχυθεί το προσωπικό του γραφείου του και σε άλλες πόλεις αποκεντρωμένα και ιδιαίτερα στην Τούσλα. Η Ομοσπονδία δεν ε, περιορίζεται μόνο στο Σαράγεβο. Και στο Μόστα, και στην Τούσλα ε, θα πρέπει να έχουμε εκπροσώπους του γραφείου μας. Και σε σχέση με τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και τους βιασμούς θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή στη Βοσνία Ζεγοβίνη εκδίδονται καταδικαστικές αποφάσεις κατά των εγκλημάτων πολέμου αυτών των, βιαστών. Αλλά δεν αποζημιώνονται τα θύματα, τιμωρούνται με ενηθίτες, αλλά δεν υπάρχει καμία αποζημίωση ούτε ηθική ούτε ηλική. Και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ασχοληθεί και να βοηθήσει τα θύματα. Γιατί εάν αρχίσουν να λύνονται μία, δύο, τρεις υποθέσεις, θα υπάρξουν δυνατότητες να βρεθούν και κονδύλια για την αποζημίωση των θυμάτων αυτών των εγκλημάτων πολέμου και την καταδίκη των, ε, εγκλημάτων. Η δική μας πολιτική ομάδα, οι φιλελεύθεροι, υποστηρίζουν λοιπόν την έκθεση και συγχαίρουν την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Thank you. <clears throat> Um, in this uh, report... Ευχαριστώ. Στην έκθεση αυτή, αυτό που νομίζω έχει καταστεί σαφές, είναι ότι το αμφιλεγόμενο σημείο είναι το κατά πόσον πρέπει να δούμε τη χώρα ως μια όρημη δημοκρατική χώρα, Ω μια κοινωνία που ακόμα είναι διχασμένη μετά από τι εχθροπραξίες. Αν θα πρέπει να αναθέσουμε περισσότερε ευθύνε στις αρχές, ώστε να υπάρχει περισσότερη ανάληψη ευθυνών σε τοπικό επίπεδο, ή αν οι στρατηγικέ μας θα πρέπει να βασίζονται σε πολύ αυστηρά κριτήρια, και αν αυτό μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την δράση των ντόπιων. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι Βρήκαμε πολύ καλέ συμβαστικέ λύσει, μεταξύ άλλων τροπολογία 4 για την κατάργηση του γραφείου τη Επατηθαρμοστία. Καθησυχάστηκαν κάποιε από τι ανησυχίε μα, αλλά υπάρχει και άλλο περιθώριο βελτιώσεων. Διότι κάποια απογοήτευση σε όλου μα συμβαίνει να γεννάται κατά καιρού. Και όσο για τη συμβαστική πρόταση για τους Βουχαμπή, νομίζω ότι είναι κάπως δυσανάλογο να αναφέρεται. Νομίζω οι θρησκευτικοί εξτρεμισμοί, οι εθνοτικοί εξτρεμισμοί σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να καταδικάζονται γιατί προκαλούν διακριτική μεταχείριση, βία, συγκρούσεις και αυτό το είδαμε στην παρέλαση, την Gay Pride στο Βελιγράδι και στο Split. Είδαμε τις αντιδράσεις που υπήρχαν σε όλη τη χώρα από καθολικούς. Όμως, το να αναφέρεται εδώ στην έκθεση για τη Βοσνία το θέμα αυτό δίνει κακή εικόνα για τη χώρα και ουσιαστικά ενοχοποιεί τους Ισλαμιστές και επίσης δίνει την ευκαιρία στο ακραίων ε, το χριστιανικό κόμμα που ασκεί διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών και των οποίων τα παιδιά δεν εμβολιάζονται για σοβαρέ ασθένειες, θανάσιμες ασθένειες λόγω των ακραίων χριστιανικών επιθέσεων, δίνει λοιπόν σε αυτό το κόμμα μια καλύτερη εικόνα. Και κάποιοι από αυτού ε, δεν είναι καλύτεροι από του μετριοπαθεί Ισλαμιστές. Ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Η Ντόρις, η Ντόρις ως συνήθως έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό κείμενο και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη και με το ίδιο το κείμενο και με τις συμβαστικές τροπολογίες. Απλώς μία παρατήρηση να κάνω και δεν θέλω να εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Η τέταρτη συμβαστική πρόταση. Νομίζω τελικά δεν βελτιώνει το αρχικό κείμενο. Το προτιμούσα. Νομίζω θα έπρεπε να αναφερθούμε στο 5 2. Αυτό είναι μια ε, λύση που θα μπορούσε να αποδεχτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είναι μια λύση, μια φόρμουλα που πάντοτε την ε, ακολουθούσαμε. Το ψηφίσμά μας θα είναι αντικείμενο ανάγνωσης πολύ προσεκτικής στην ε, περιοχή αυτή. Κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε γίζεται και μετράται, εκτιμάται πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, ό,τι και αν πούμε, τον, τον παραμικρό που θα πούμε θα τον προσέξουν πάρα πολύ στην ε, Βοσνία. Και θα μας ε, θέσουν και ερωτήματα μετά. Θα μας ρωτήσουν γιατί δεν αναφέρουμε πλέον το 5 2. Διότι το 5 2 σημαίνει ότι η διεθνή κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν και εκείνες δικαίωμα λόγου Διότι αν πλέον περιοριστούμε στις δύο απαιτήσει, αυτό μπορεί να ερμηνευτεί στη Βοσνία και να θεωρήσουν ότι μόνο δύο σημεία απομένουν να υλοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι τα πέντε υπόλοιπα έχουν ήδη διευθετηθεί. Νομίζω λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουμε στο αρχικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μπορούμε στις εκθέσεις μας να σημειώνουμε και τα θετικά. Ο κύριος ε, Βάγγελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα λίγο να επανέλθω σε ένα θέμα της σημερινής συζήτησης που θεωρείται λεπτομέρεια. Θέλω να υποστηρίξω πάρα πολύ ηθικά την εισηγήτρια, την κυρία Ντόρις Πακ. την κοινή γνώμη, ε, διάφορα μέσα ενημέρωση στη Βοσνία κάνουν μια εκστρατεία και πρέπει να αναφερθώ σε αυτό γιατί έχουμε σήμερα εκπροσώπους και των μέσων ενημέρωσης και του πολιτικού κόσμου της Βοσνίας σερσεχοβινης Εμείς είμαστε δημοκρατική κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι όσοι συζητούν για το δημοκρατικό ευρωπαϊκό μέλλον ε, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης εύχονται στη χώρα αυτή ε, όσο γίνεται να είναι ε, απρόσκοπτη η ευρωπαϊκή της πορεία. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχθούμε οι δικοί μας εισηγητές και τα μέλη του Κοινοβουλίου να αναμειγνύονται, να προσπαθούν να τους αναμειγνύουν ε, στην εσωτερική πολιτική συζήτηση με τρόπο απαράδεκτο. Αυτό συμβαίνει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, αν θέλουμε να έχουμε καλή συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κοινή γνώμης ε, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και να πω και ένα δεύτερο. πιστεύω όντως ότι δεν είναι απαραίτητο να υπερτονίζουμε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή ένα σημείο. Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές θρησκευτικέ κοινότητες. Η Βοσνία, Ερζεγοβίνη, είναι ένα κράτος ε, ακριβώς πολυσυλλεκτικό για ε, τη συνύπαρξη Ε, και έγινε και πόλεμος μεταξύ των κοινοτήτων. Τώρα έχει τελειώσει βέβαια, αλλά ε, παραμένουν οι διαφορές. Θα, δεν θα πρέπει να τονίζουμε υπερβολικά κάποια φαινόμενα στα κείμενά μας. Εγώ θα ήθελα να αποφύγω αναφορά στους Ουαχαμπίτες. Δεν χρειάζεται να το τονίσουμε τόσο πολύ. Δεν είναι χαρακτηριστικό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ούτε του μέλλοντός της. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή που είναι πάρα πολύ ισορροπημένη και για τις προσπάθειές της, καθώς επίσης και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Για να ανοίξουμε όλες τις προοπτικές στη Βοσνία Ζεγοβίνη ε, όταν υλοποιηθούν ε, οι προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η μακρά πείρα τη εισηγήτριας και η πολύ κοντινή γνώση των όσων συμβαίνουν στη χώρα. Είναι πράγματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε από το ίδιο το κείμενο του ψηφίσματος. Η εισηγήτρια περιγράφει τα προβλήματα ακριβώς ως έχουν, χωρίς να υπερβάλλει ούτε να τα υποβαθμίζει και μαζί με τους κοιόδης εισηγητές κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τη χώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν, υποκρύπτονται καλές προθέσεις εδώ. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Πάκ λοιπόν για αυτή την έκθεση. Ξέρω ότι έχει τη συνήθεια να δέχεται, έχει συνηθίσει να δέχεται συγχαρητήρια, αλλά από καιρούς καιρών δεν κάνει κακό να επαναλαμβάνει κανείς τέτοιες συνήθειες. Το ίδιο το ψήφισμα. δίνει μια ευκαιρία να δώσουμε μια όθηση για κάποιες θετικές εξέλιξεις στη Βοσνία-Ριζεγοβίνη παρόλο που στις περισσότερους τομείς υπήρξε περιορισμένη πρόοδος στην πορεία για την ευρωπαϊκή ένταξη, νομίζω ότι με την πρόσφατη κυβέρνηση δεν θα υπάρχουν πλέον δικαιολογίε για άλλες αναβολές και για μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Η Βοσνία Ριζεγοβίνη θα πρέπει να αναπτύξει μια κουλτούρα συμβιβασμού και επικοδομητικού διαλόγου, κάτι που θα είναι η βάση, η απαραίτητη βάση, τα θεμέλια για όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Για τους κρατικούς νόμους και την άρση των λογοκρισιών, αυτό δείχνει ότι η χώρα μπορεί να επιτελέσει θετική πρόοδο. Θα μπορέσει να χειριστεί την ευρωπαϊκή της πορεία και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρξει ευρεία πολιτική συμφωνία για ουσιώδη ζητήματα και αν υπάρξουν ε, θεσμικά όργανα που να λειτουργούν εύρυθμα σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. Νομίζω ότι οι ιδέε που απηχούνται στι περισσότερε τροπολογίε είναι μια πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε με την πορεία και τι μεταρρυθμίσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και τι στηρίζω τι συμβαστικέ τροπολογίε, ιδίω αυτές που αναφέρονται στα φαινόμενα του εξτρεμισμού ή στο γραφείο του ΙΠΑ του Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη να προχωρήσει στη διαδικασία ένταξης. Και αυτό για να υπάρξει ταχύτερη εξέλιξη της χώρας και για την ίδια την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, αλλά κατά κύριο λόγο προς όφελος των ίδιων των πολιτών της χώρας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χάσαμε το βιβλίο τη αντιπροσωπεία, αλλά δεν πειράζει. Είναι ευχάριστο να κατηγορήσω την παρούσα θέση. συγγνώμη που καθυστέρησα. Ευχαριστώ του συναδέλφου, Κάτσεν και Φάγγελ, οι οποίοι ε, μίλησαν για του φιλελευθέρου. Με ισχυώδη εισηγήτρια, οπότε να ευχαριστήσω την Τόρι Πακ, μια που νομίζω ότι κατέληξε σε αυτή την πάρα πολύ καλά ζυγισμένη έκθεση. Έχουμε τη συμβαστική 4, επί της οποίας πιστεύω το εξή ότι, κοιτάξτε, τα συζητήσαμε για το 5 συν και για ε, πάμε πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά να αναφέρονται, αλλά ήθελα να επισύρω την προσοχή σας σε... Ε, στο πόσο αποτελεσματική είναι η διατύπωση του 4, εκεί που αναφέρει την διάλυση της Βοσνίας Αζεγοβίνης. Λέει όμως ότι οι αρχές της χώρας θα πρέπει να επιλύσουν κλπ. λοιπά. Επομένως, είναι σαφής η σχέση, ο σύνδεσμος μεταξύ του ενός και του άλλου. Άρα θέλουμε να υπάρχει τέτοιου είδους αποτελεσματική διατύπωση. Επίσης, όσον αφορά την συμβαστική 8, προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε την κατάσταση αυτή με τους Βαχαμπίτες και είπαμε ότι καταδικάζουμε πάσα ακραία πολιτική τάση και εξτρεμισμό. Επομένως, αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι ναι, έχουμε πολλές ακραίες τάσεις, οι περισσότερες από τις οποίες ε, έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία της χώρας. Και είπαμε ότι ο Ουαχαμπισμός έχει εισαχθεί στη χώρα. Άρα αυτό που μας θέλουμε να να υπόψη ότι υπάρχει αυτή η ε, γενική κάθετη αντίθεση σε κάθε εξτρεμισμό που πρεσβεύει το μίσος και τη χρήση Στο 45 τώρα. Επ' αυτού θεωρούμε ότι θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο το πόσο χρειάζονται κάποιες μεταρρυθμίσεις μετά από διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, με πλατφόρμα κάποια διάσκεψη κλπ. Άρα θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα βολέψουμε το 45 τελικά. Uh, Και εγώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την Doris Πακ ε, για τόσο καλά τεκμηριωμένη έκθεση και τα είπε ο σκιώδης πολύ καλά, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως για τους Βαχαμπίτες. Νομίζω ότι καλά τα λέει η συμβαστική 8 Αλλά θα πρέπει να προβληματιστούμε. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτή την περιοχή, αφορά όλο τον κόσμο. Στην οδιακτή της Μεσογείου και στις ίδιες τις χώρες μας έχει εξαπλαθεί. Και πιο βλέπω εκτός Αδικής Αραβίας βρίσκονται στο Λονδίνο. Βελγκρέβια, Νότια Προάστια κλπ. Επομένως, να. Πώς εξάγει το καθεστώς Σαουδικής Αραβίας αυτόν τον εκτρεμισμό; Άρα θα πρέπει να το συζητήσουμε. Πώ γίνεται αυτή η εξάγωγη λοιπόν των Οχαμπιτών σε όλο τον κόσμο, και στη Συρία. Άλλωστε συμβαίνει το ίδιο. Επομένω, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την Doris Πακ. Κύριε κυρία Πακ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ο στόχος μου δεν ήταν τώρα να συζητάμε όλες ολόκληρες για τους Ουαχαμπίτες. Έπρεπε να το πω όμως γιατί κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωση στη Βοσνία και με λάθος τρόπο. Και αυτά τα λάθος που είπαν πρέπει να τα συζητήσουμε. Και πάλι στα γερμανικά έχουμε μια παροιμία που λέει ε, ότι θα πρέπει να ε, πνιγεί ε, το κακό στη ρίζα του. Είναι μεγάλη η Ισλαμική κοινότητα στη Βοσνία και αν ριζώσει αυτό το κίνημα ε, του αγαπητισμού, θα έχουμε πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το υποτιμούμε και να το θεωρούμε λεπτομέρεια. Θα πρέπει να το κατονομάζουμε, αλλά ε, μαζί με άλλες εξτρεμιστικές και εθνικιστικές συμπεριφορές και εκφάνσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι βρήκαμε μια πολύ καλή διατύπωση. Εγώ δεν κατηγορώ τη Βοσνία, ε, προειδοποιώ για ένα κίνδυνο που δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθός του. Εάν δεν του βάλουμε φρένο τώρα στη ρίζα του, στην αρχή του, ε, θα το μετανιώσουμε. Πόσα χρόνια, τα, ε, τα τελευταία 20 χρόνια, πόσες φορές έχουμε πει στενή μου γνώση να σήγα πρώτα. Γι' αυτό έτσι ήθελα να το συζητήσουμε χωρίς ε, αρνητική φόρτιση. Είναι καλό αυτό που κάνουμε, δεν είναι κακό. Ε, είναι ε, στραμμένη στο μέλλον. Τι δουλειά έχει η Σρεμπρένιτσα, γιατί το συγκρίνουμε. Ανέκαθεν την έχουμε καταδικάσει αυτή την κατάσταση, επίσης καταδικάζουμε εκείνους που την αρνούν. Δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, τα κατονομάζουμε και καμιά δουλειά δεν έχουμε να κατέβουμε ανώμια πράγματα. Είπε ο κύριος Κατσίν, ότι θέλω να φύγει ο ύπατος εκπρόσωπος. Ναι, αλλά είμαι η συγγήτρια του Κοινοβουλίου και έχω ένα κείμενο έκθεσης για όλο το Κοινοβούλιο και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Έχω τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Η κυρία Μποσκούρτ δεν συμφωνεί με το συμβιβασμό, δεν είναι ικανοποιημένη για τα μεθοριακά ζητήματα. Βέβαια λέει θα το ψηφίσει. Έχει κάνει μια τροπολογία η κυρία Μποσκούρτ που για παράδειγμα αναφέρεται στον κύριο Γιωσίποβιτς, Κροάτι Πρόεδρο, και τι είπε για τις αλλαγές των συνόρων. Τι δουλειά έχουν αυτά τα κείμενα στη συγκεκριμένη έκθεση. Δεν θα πάω να πω τι είπε κύριο Τάντιτ ή ο άλλο γείτονα πρόεδρο για τη Βοσνία. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η Βοσνία Ερζεκοβίνη. Και παρακαλώ να βρούνε λύσει με του γείτονέ του. Και όταν συζητήσουμε για την Κροατία με το καλό στην έκθεση της Κροατίας, τότε θα αναφερθούμε στον πρόεδρο της χώρας. Είπε το Α, το Β, προσβλέπουμε κτλ. Ε, παρακαλώ αυτή την τροπολογία της κυρίας Μινέμπο Κούρτ να μην τη δεχτούμε, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει καμιά δουλειά να αναφέρει η έκθεσή μας πρόεδρο γειτονική χώρας. Αυτά. Τώρα, άλλη ιστορία που λίγο, πώς να το πω, με βαραίνει πάρα πολύ. Καλό θα ήταν ε, αν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό πρότεινε ο κύριος Κάτσιν και λίγο η κυρία Λάτφορτ το επενήχθηκε. Οι συνάδελφοι φιλελεύθεροι επιθυμούν να διοργανώσουμε διεθνή διάσκεψη όπου να ξανασυζητήσουμε τον Dayton με τους ενδιαφερομένους, επιτόπου, ενεχομένους κτλ. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει μαζί με τα ξερά να κάψουμε και τα χλωρά. Τρομάξαμε να βρούμε κυβέρνηση, πώς το λένε τώρα αυτό, Υπουργικό Συμβούλιο. Ε, και έχουν ε, νόμους που πρέπει να υλοποιηθούν και μόλις εγκρίθηκαν. Τώρα λοιπόν που αρχίζει λίγο να αποκτά μια κρατική υπόσταση το κράτος, δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς έξωθεν ότι, α, κοιτάξτε, τώρα χρειαζόμαστε διεθνή διάσκεψη για να εξετάσει τον Dayton. Αυτό είναι τελείω αντιπαραγωγικό. Δεν γίνεται ανταπαραγωγικότερο. Εμεί δεν είμαστε δάσκαλοι που θα του δασκαλέψουμε. Θέλουμε να του βοηθήσουμε. Οι άνθρωποι επιτόπου θα πρέπει να το καταλάβουν και οι πολιτικοί επιτόπου τώρα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Προσπαθούν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα και στην περίπτωση Φίντσι που γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει μια απόφαση που πρέπει να υλοποιηθεί. Αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο στο ιστορικό της χώρας. Βεβαίως με τη βοήθειά μας εφόσον την επιθυμούν. Αλλά τώρα να διοργανώσουμε και πάλι διεθνή διάσκεψη. Θυμηθείτε την τελευταία ε, ε, που απέτυχε ικτρά προσοχή να βοηθήσουμε τον κόσμο αλλά να του αφήσουμε να αναλάβουν τις τύχες τους και τις μοίρες του. Και όσο ε, ε, γρηγορότερα μπορεί να φύγει ο ύπατος εκπρόσωπος, τόσο καλύτερο. Γιατί αναλαμβάνουν εκείνοι τις ευθύνες και δεν τις παραπέμπουν σε αυτόν. Συγγνώμη που φορτίζομαι συναισθηματικά. Ξέρετε ότι το θέμα με συγκινεί και με ενδιαφέρει. Δεν θα πρέπει να είμαστε πάντα οι δάσκαλοι όλων των εθνών. Να είμαστε ε, ευαίσθητοι και όταν εγώ λέω ευαίσθητοι το εννοώ. Θα πρέπει να μάθουμε όλοι και μάθαμε και στα Βαλκάνια ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στις ευαισθησίες του κόσμου. Στη Βοσνία Ζεγοβίνη δεν θα το κάνουμε αν αρχίσουμε να τις κουνάμε το δάχτυλο θέλουμε διεθνή διάσκεψη. Και ε, ο πρώτος που θα αντιδράσει θα είναι ο Ντόντιφ και πάλι θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας εδώ και χρόνια ε, το συζητάμε, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ελπίζω αύριο να ψηφίσετε όλοι. Έχω κάνει ένα πάρα πολύ καλό κατάλογο ψηφοφορία. Μη φύγετε, λέει ο Πρόεδρο, ε, λέει κάποιο το λόγο. Ε, η, κυρία Λούνατσεκ για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που απειλείται όμως πρέπει να πάει να ψηφίσει η κυρία Πακ. Δεν άκουγα τι λέγατε, Πρόεδρε. Πρέπει να φύγει η κυρία Πακ, έλεγα. Εντάξει, Ντόρι, συγγνώμη, που ζητώ το λόγο, θα πρέπει να διαφωνήσω σε ένα σημείο. Προσπάθησαν οι πράσινοι ε, αυτό το θέμα με τους Ουαχαμπίτες να το βάλουν αλλιώς ε, στη συμβαστική πρόταση για να ε, καταδικάσουμε οποιαδήποτε εξτρεμιστική και ακραία έκφραση, όχι μόνο αυτή. Ήθελα να το διευκρινίσω μόνο. Is... Μάλιστα. Ολοκληρώνεται εδώ αυτό το σημείο της ημέρησης διάταξης. Ευχαριστώ πολύ, Ντόρις. Πριν περάσουμε στο επόμενο που είναι η Τουρκία... Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Θεοχάρους για μια σύντομη δήλωση. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Thank you for giving me the opportunity to present the... Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο και ανθρωπιστικό που ε, περίλθε στη γνώση μου εχθές το βράδυ. Γνωρίζετε ίσως ότι ο τουρκικός τύπος πρόσφατα ε, είχε πολλά δημοσιεύματα που ενδιέφεραν ε, τον κόσμο. Στη φυλακή του Διαρμπακύρ βρέθηκαν 38 σκελετοί σε μια διαδικασία κανονική ανακαίνησης και τα κρανία ε, όλα φέρουν τραύμα οποίοι από σφαίρα περιστρόφου 9 χιλιοστών. Αυτά τα έχουμε δει και στην Κύπρο ε, στους ομαδικούς τάφους. Τα λείψαν αυτά, ε, ελέγχονται ε, με DNA και διαδικασία και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με αγνοομένους Τούρκους ή Κούρδους. Ζητώ λοιπόν την υποστήριξη της ομάδας και του της Επιτροπής συγγνώμη, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε ε, οι επιστημονικοί φορείς ε, της Κύπρου να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα λείψανα. Γιατί εκατοντάδες οικογενειών ζουν μια ε, τρομακτική αγωνία στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες πάνω από 200 αγνοούμενοι μετά τον πόλεμο του 1974 ήταν κρατούμενοι στις φυλακές του Διαρμπακίρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Θα πρότεινα να απευθυνθούμε στην τουρκική πρεσβεία και να παρακαλέσουμε να διευκρινιστεί. Και με την κυρία εισηγήτρια στη συνέχεια να το συζητήσουμε, τι δρόμο μπορούμε να βρούμε ε, για να το διευκρινίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Επόμενο σημείο λοιπόν, Τουρκία. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια μας, την κυρία Όμεν Ράιτεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, στις 12 Ιανουαρίου εδώ στην Επιτροπή μας κατέθεσα το σχέδιο ψηφίσματος για την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας. Ήδη από τότε είχα πει ότι θέλω τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μάλλον τη συμμερίζομαι όπως και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι η Τουρκία παίζει ρόλο κλειδί ως χώρα για την ασφάλεια και για την ευημερία πλέον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στο σχέδιο ψηφίσματός μου αναφέρω την αλληλεξάρτηση ε, της Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το πράττω αυτό. Υπάρχει το έδαφος για οικονομική ανάπτυξη στην Τουρκία και επίση έχει σημαντικό ρόλο η Τουρκία για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό και τις δυνατότητες συνεργασίας και συνέργειας. Το έχετε και εσείς πει, Πρόεδρε, στην εξωτερική πολιτική ε, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Λοιπόν, έχουμε αμοιβαία εξάρτηση ε, με θετικά αποτελέσματα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Τουρκία. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να υπάρχουν και αμοιβαίε συνεννοήσεις. Τι σημαίνει αυτό. Ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Τουρκία οπωσδήποτε θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να ανταποκριθούν σε αυτές τις δεσμεύσει τους. Για την Τουρκία είναι συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων που περιμένουμε, αλλά όχι μόνο αυτό θα πρέπει να υπάρξει και βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με τους γείτονές της. Εγώ περιμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της υποστήριξη για τη νέα ατζέντα του Επιτρόπου Φύλε για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Περιμένω όμως επίσης και νέες ε, προσπάθειες για να δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις να προχωρήσουν ορισμένα κεφάλαια. Θα επανέλθω σε αυτό, Πρόεδρε, και για τις μεταρρυθμίσεις ε, και στη δικαιοσύνη και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι απαραίτητο να το τονίσουμε αυτό. Και στην εξωτερική πολιτική, Πρόεδρε, κατά πολέμηση τρομοκρατίας, Φερρυπίν, μπορούμε, εάν εργαστούμε από κοινού και πιο στενά, να έχουμε αποτελέσματα και στην Ένωση και στην Τουρκία. Πρόεδρε, ήδη από το Γενάρη εξέφρασα τη μεγάλη μου ανησυχία για την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθεροτυπία, ε, για την προφυλάκηση που διαρκεί τόσο πολύ και τις τόσες ε, συλλήψεις ε, ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών, δημοσιογράφων. Αυτό το μήνυμα το υποστήριξαν και οι συνάδελφοί μου εδώ παρόντες και τα μέλη της Επιτροπής και τους ευχαριστώ. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι ότι τώρα περισσότερο από ποτέ έχει σημασία να έχουμε μια στεναρή, ε, ισορροπημένη αλλά και αντικειμενική θεώρηση και ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα ε, που να μπορούν να το εξεργαστούν και να το αξιοποιήσουν. Τι εννοώ, ότι δεν μπορούμε όλες τις λεπτομέρειες και τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους να τα βάζουμε σε όλα τα ψηφίσματα. Αν κάθε χρόνο βάζουμε ε, στα ψηφίσματά μας ε, ε, ακόμα ένα θέμα, θα φορτωθούν πάρα πολύ. Λοιπόν, έγινε συζήτηση τον Ιανουάριο. Έχουν κατατεθεί 461 τροπολογίες στη εβδομάδα του Στρασβούργου θα αναζητήσω συμβαστικές με τους συναδέλφους. Τους ευχαριστώ για τη συνεργασία τους. Είναι πάρα πολύ επικοδομητική πάντα και καλή. 29 ε, είναι οι τροπολογίες αυτές, οι συμβιβαστικές, ε, που ε, εστάλησαν τη Δευτέρα το βράδυ, αργά βέβαια, πολύ αργά σε κάθε συμβαστική ε, τροπολογία υπάρχει ένα μήνυμα κλειδί. Αυτό που δεν έκανα εγώ στο σχέδιο έκθεσης ήταν το εξή, Μάλλον το πω Ανέφερα τον αντιτρομοκρατικό νόμο ε, ότι οδήγησε σε πολλές συλλήψεις και κρατήσεις και προφυλακίσεις, αλλά αυτό που δεν είχα κάνει ήταν να αναφέρω συγκεκριμένα ε, στοιχεία. Τώρα στους συμβιβασμούς αυτό το έχουμε κάνει είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι ε, για την αντιτρομοκρατική ε, νομοθεσία και το ποινικό κώδικα. Γιατί ε, οι ορισμοί έχουν πολύ ευρία ερμηνεία και εφαρμογή. Τώρα αναφέρουμε συγκεκριμένα άρθρα των νόμων που επιγόντως θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Ένα άλλο σημείο που ήρθε πολύ συχνά στη συζήτηση ήταν η σχέση κυβέρνηση αντιπολίτευσης. Τονίζω πάντα με τους συναδέλφους ...τις συμβαστικές τροπολογίες τη σημασία του διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και συνεργασίας πάντα. Εκφράζουμε και τη μεγάλη μας ανησυχία για τις ε, δίκες που εκκρεμούν ε, κατά ε, μελών του τουρκικού κοινοβουλίου της μεγάλης τουρκικής εθνοσυνέλευσης και αρχηγού μεγάλου κόμματος της αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί οι βουλευτές να λειτουργούν υπό την απειλή της ποινική δίωξης. Αυτό δεν συνάδει ούτε με τη δημοκρατία ούτε με την ελευθερία της έκφρασης των βουλευτών και των πολιτικών. Και ε, κάτι άλλο ακόμα που διευκρινίσαμε ήταν η ιστορία του Χραντ Ντίνκ. Ε, η απόφαση δικαστική ήταν απογοητευτική. Και για μένα αυτή η δίκη είναι η δοκιμή ακριβώς ε, που θα κριθεί αν λειτουργεί καλά το κράτος δικαίου, κατά πόσο είναι ανεξάρτητη και ακομάτιστη η δικαιοσύνη στην Τουρκία. Και τώρα τι γίνεται. Το τονίζουμε και φέτος, όπως και τα προηγούμενα έτη, ότι θα πρέπει να γίνει πραγματική διερεύνηση ε, της υπόθεσης ε, της δολοφονίας του Χραντ Ντίνγκ και ε, να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης ε, ε, όλοι οι υπεύθυνοι και οι αυτούργοι και όχι μόνο οι αχυράνθρωποι τους. Επίσης, κάποιες άλλες προσαρμογές η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών καλωσορίζουμε ως πρώτο βήμα, πρώτο βήμα τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνη, αλλά ε, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κοιτάξει τι βήματα ε, χρειάζονται να γίνουν για να ανοίξει το κεφάλαιο 24. Πρόεδρε, είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν έχω το χρόνο, καταλαβαίνω από εσά να μπω σε λεπτομέρειες. Ε, διαβάζοντας όλα αυτά ε, που λένε οι συμβαστικές ε, τροπολογίες θα τα καταλάβουν οι συνάδελφοι. Έρχομαι τώρα στην Κύπρο, Πρόεδρε. Ένα σημείο όπου δεν καταφέραμε να κάνουμε συμβαστική τροπολογία. Και για ποιο λόγο. Διότι το κείμενο στο σχέδιο ψηφίσματος δεν είναι απλώς αντικειμενικό, αλλά είναι πάρα πολύ προσεκτικό και πολύ συγκεκριμένα γράφει ποιο είναι το μήνυμά μας για τις σχέσεις Τουρκίας-Κύπρου. Και θα παρακαλούσα όλους τους συναδέλφους όλες τις τροπολογίες που έχουν σχέση με την Κύπρο ε, να τις κοιτάξουν. Αν θέλετε μπορείτε να τις αποσύρετε ή να τις αφήσετε να ε, τις ψηφίσουμε, αλλά εγώ εμένω στο δικό μου κείμενο. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε, όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτή την προσπάθεια και ελπίζω αύριο να πάει καλά η ψηφοφορία. διευκρινίζει τα πράγματα αυτό το ψήφισμα, ξεκαθαρίζει αλλά και διατρανώνει κάποια άλλα και νομίζω ότι είναι πολύ καλό και μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος, Thank you, Mr. Chairman, and thank... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την Ρία, την ε, εισηγήτρια. Εξαιρετικό το έργο το οποίο επετέλεσε. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σωσμένη, πάρα πολύ θετική. Ακριβώ και όπω είναι και θετικά και τα όσα προτείνει ο Επίτροπο Φούλερου, ούτω ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα πρόοδο σε σχέση με την Τουρκία. Ε, η δική μα πολιτική ομάδα έχει ουσιαστικά βοηθήσει μέσω των τροπολογιών και όσον αφορά τι διαπραγματεύσει με τη Ρία. Για να καταλήξουμε σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα γιατί είναι ό,τι, ό,τι χρειάζεται αυτό για τον ε, στόχο μας μια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να κοιτάξουμε τις ε, σχέσεις μας με την Τουρκία, τώρα που περισσότερο από ποτέ, είναι πιο σημαντική. Είναι σημαντική για την ευρύτερη περιοχή. Με θετικό τρόπο. Πάντως έχουμε εδώ και κάποιες νέες προκλήσεις. Από τον Ιούλιο θα έχουμε την Κύπρο στην Προεδρία της Ένωσης. Και οπωσδήποτε αυτό πρόκειται να απαιτήσει προσοχή από κάθε πλευρά και σίγουρα από την τουρκική πλευρά σε σχέση με το τι μορφή θα λάβουν οι σχέσεις με την Ένωση. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέει έκθεση όσον αφορά το άνοιγμα των νέων κεφαλαίων, 23-24. Και επίσης η δυναμική αυτή, η διατύπωση. Εκεί να φαίνονται τα πιο σημαντικά των προβλημάτων. Δικαιοσύνη, δηλαδή. And uh, uh, of course in the lack or in the problems. Βεβαίως και τα θέματα σε σχέση με πλουραλισμό στα ΜΜΕ, αλλά και την ελευθερία της έκφραση γενικότερα. Ε, φυσικά έχει σημασία και η διερεύνηση των συνδικών θανάτων του Χραντίνγκ και πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εντρογνωτική νομοθεσία πώς ε, χρησιμοποιείται για καταστολή ε, αντιπολίτευσης ε, φημώματος των φωνών διαφωνίας τέλος πάντων για την Κύπρο, η δική μας πολιτική ομάδα επιθυμεί να υπάρξει μια δίκαιη ρύθμιση. Θα διευκολύνουμε επομένω οποιοδήποτε τρόπο διαλέξουμε για να πάμε προς αυτό το αποτέλεσμα και πρέπει να θυμίσουμε ότι χθες είχαμε επαφές με το Συμβούλιο. Τους ρώτησα Τι λένε για αυτή τη διάσκεψη με την Συρία που θέλει να οργανώσει η Τουρκία. Βέβαια θα κληθεί και η Κύπρος εκεί ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεώρησε επομένω ότι το ζήτημα αυτό πρόκειται να καλυφθεί αποτελεσματικά από την έκθεση. Και πάλι σε συγχαρητήρια από την υπόλοιπη μας ομάδα προς την εισηγήτρια. Επίσης, ε, εκ μέρους του κύριου Μπιόρς, του Σιώδους εισηγητού μας, ε, να σου πω ότι και εκείνος ε, ευχαριστεί, συγχαίρει. Δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω λέει κύριο Λάμστροφτήρια Όμεν Ρόιτεν για την καλή τη εργασία. Εδώ και μήνες, ένα χρόνο περίπου, ε, συμφωνούμε ότι η κατάσταση έχει το εξή παράδοξο. Διαπραγματεύσεις ενταξιακέ έχουμε με την Τουρκία. Κανονικά αυτό θα πρέπει να ήταν θετικό. Και αυτό οδήγησε στο ότι έχουμε δυσκολίες σε άλλου τομείς της συνεργασίας, ιδιαίτερα στο στρατηγικό διάλογο για την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό θεωρώ πολύ καλό που έχουμε μια θετική ατζέντα πλέον που δεν επικεντρώνεται, δεν ε, έχει μια αιμονή ε, στην προεταξιακή διαδικασία, δεν την υποτιμά, αλλά δεν δυσκολεύει την υπόλοιπη συνεργασία. Η έκθεση έχει δύο σημαντικά μηνύματα. Πρώτον, είναι επικριτική για τα βασικά θέματα που μας ενδιαφέρουν και ως ομάδα. Ε, ανθρώπινα δικαιώματα, βασικές ελευθερίες, κράτος δικαίου και δημοκρατία. Η Τουρκία ως υποψήφια χώρα θα πρέπει να αποδείξει την προθυμία της ε, να ανταποκριθεί ε, και μάλιστα διαρκώς, όχι στιγμία και μεμονωμένα κατά καιρού. Επίσης διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται ε, σημαντικά σε κάποιους τομείς και μας ανησυχεί. Το Δεκέμβρη δεκάδες δημοσιογράφοι συνελήφθησαν και κρατούνται ακόμα στις φυλακές. Αυτό είναι απαράδεκτο. Στο παρελθόν χαιρετήσαμε τα ανοίγματα της κυβέρνησης προς τους Κούρδους. Τώρα ανησυχούμε γιατί επιδεινώνεται και η κατάσταση. Θα πρέπει να πω όμως το εξή ξεκάθαρα. Εάν θέλουμε ειρηνική επίλυση του Κουρδικού στην Τουρκία, θα πρέπει αυτό να το επιδιώκουν όλες οι πλευρές. Από ε, ε, την ε, σύλληψη του Τσαλάν ε, έχουν δεχτεί επιθέσεις ε, ε, σε πολλές χώρες και πολλές πόλεις και στην εκλογική μου περιφέρεια γραφεία εφημερίδων και μέσων ενημέρωσης. και πήγα και εγώ και τους επισκέφθηκα και το ξέρει και η Ρία. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Επίσης η δικαιοσύνη δεν ανταποκρίνεται στις δικές μας προϋποθέσεις. Η υπόθεση Εργένεκον μας ανησυχεί πολύ και Παρακαλώ κοιτάξτε προσεκτικά στην Κομισιόν την ε, συμβαστική 10. 11, συγγνώμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιπολαιότητα αναλύει την κατάσταση. Και με βάση το κατηγορητήριο όταν ρωτήσαμε σε μια επιστολή ε, τι λέει το κατηγορητήριο, μα απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι άμα κάτσουμε να τα αναλύσουμε αυτά, υποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη τη Τουρκία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο να το αναλύετε και να το λέτε και στο Κοινοβούλιο. Η συνταγματική μεταρρύθμιση. Ε, συνεργαζόμαστε στη μεικτή Κοινοβουλευτική με την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, αλλά το 2010 ήδη υπήρξε αναθεώρηση του συντάγματος και πού είναι η υλοποίηση ε, των όσων αποφασίστηκαν στη συμβαστική 5 ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την ε, λεπτομερή παρατήρηση να την ε, περιγράψει σε μια λεπτομερή έκθεση γιατί πώς έχει η κατάσταση. Ανησυχούν πάρα πολύ οι συνομιλητές μας στην Τουρκία. Αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνούμε ότι τα κεφάλαια 23 και 24 θα πρέπει το συντομότερο να ανοίξουν. Θέλουμε τη θετική ατζέντα, τονίζουμε το στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο στρατηγικός διάλογος πρέπει να συνεχιστεί και Χαίρομαι που είναι κάποιος από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση παρόν για να μιλήσει ε, και είναι σημαντικό και να δείξουμε και στου Τούρκου ε, φίλους μας πόσο σημαντική είναι η θέση τους για την εξωτερική πολιτική και της Ένωσης. Και ένα τελευταίο. Τι μέλη γενέστε. Θα ήθελα κάποιες πρόοδο στο θέμα της ε, θεώρησης διαβατηρίων και της απελευθέρωσης, γιατί μετά την Τελωνιακή Ένωση γίνεται αυτή η συζήτηση. Ελπίζω να βοηθήσει αυτό για θετικές εξελίξεις στις σχέσεις μας ε, με την Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Αυτό που είπατε τώρα κύριε Λάμστορφ, ανάλυση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας υποστηρίζω ρητά και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημά μας. Έχει και καθήκον νομίζω να αναλύει την κατάσταση και να συνεργάζεται και από πλευρά διοικητική ε, και να βοηθάει την νομοθετική ε, πτυχή του Κοινοβουλίου. Κύριε Φλότρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Νομίζω ότι το έργο που μα παρουσιάσετε σήμερα προ συζήτηση και για την προφορία αύριο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Πολύ ακριβή η έκθεση και πολύ σημαντική. Βέβαια κρίσιμη, αλλά νομίζω ότι η επικριτική στάση που τηρεί είναι πολύ σημαντική. Γιατί υπολογίζει τι δυνατότητε των τουρκικών αρχών να ξεπεράσουν τι δυσκολίε τι δυσκολίε, λόγω χάρη με, με τις διαδοχικές δέσμες μέτρων μεταρρύθμιση του δικουστικού συστήματο για την ελευθερία τη έκφραση, είναι μια επί... ένα επικριτικό σχόλιο αυτό πολύ συγκεκριμένο. Και νομίζω ότι μπορεί να δώσει όθηση στις τουρκικές αρχές διότι τους δείχνει συγκεκριμένους δρόμους, συγκεκριμένες ιδέες για να προοδεύσουν. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν τόσο στον τομέα των ε, θεσμικών διαδικασιών όπως και στην ε, αναθεώρηση του ποινικού κώδικα ή του νόμου κατά της θερμοκρατίας. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή πραγματικά είναι πολύ ε, καλά διαρθωμένη γιατί αναφέρεται και στις δικές μας ευθύνες ως Ευρώπης, ως Ευρωπαίων, διότι αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και να παραμείνει μια κινητήρια δύναμη για, την, ε, για τον εξυγχρονισμό της χώρας αυτής, θα πρέπει από την ευρωπαϊκή πλευρά να εφαρμόσουμε κι εμείς τις δυνατότητες δράσης που έχουμε, ανοίγοντας λόγω χάρη το κεφάλαιο 23-24 για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι η γενική προσέγγιση είναι άκρω ενδιαφέρουσα και θα έλεγα ότι η έκθεση αυτή συνδυάζεται και συμπληρώνει πολύ σωστά τη στατηγική που επελέγει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων θετικό. Δηλαδή η έκθεση αυτή πραγματικά είναι, δίνει την, τη σωστή, το σωστό έναυσμα. Δίνει ιδέες και αφετηρίες για τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στον εξυγχρονισμό και την πρόοδο της Τουρκίας. Ευχαριστώ ξανά λοιπόν την κυρία Ομερόιτεν για το ιδιαίτερα ενδιαφέρον έργο της. Θα ήθελα τώρα, επειδή με τους συναδέλφους, θα υποβλ... μαζί με άλλους συναδέλφους θα υποβάλουμε από κοινού μια τροπολογία που δεν αποτελεί μέρος των συνεργαστικών προτάσεων. Θα ήθελα να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πηγές ανησυχίε για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και οικολογικό και αρχαιολογικό αντίκτυπο ε, του τρόπου που αναπτύσσεται η Τουρκία. Δηλαδή να του πούμε προσοχή στο πώς επιλέγετε να αναπτυχθείτε, να εξελιχθείτε. Μπορεί να πληγεί η εξαιρετική, κατά τα άλλα πρέπει να το πούμε αυτό, ποιότητα του περιβάλλοντος στην Τουρκία. Νομίζω ότι και χρήσιμο θα ήταν και θα, ε, θα ακουστεί αυτό στην Τουρκία, θα περάσει το μήνυμα, εάν υποθεί κάτι τέτοιο και εγκριθεί με μια θετική ψήφο ε, μέσω τροπολογία. Νομίζω η όλη διαδικασία αυτή είναι συμβολική και εμβληματική, διότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που λένε μάλλον η δολοφονία του δημοσιογράφου Χραντίνκ έχει να κάνει με τέτοια δίκτυα και διαπλεκόμενα συμφέροντα που τελικά ε, μπορεί να κάνει τις ε, τουρκικές αρχές να αφυπνιστούν με τεκμηριωμένα στοιχεία που λένε ότι από αδράνεια δεν μπορούν να φεθούν ατιμόρυτοι αυτοργοί της δολοφονίας του Χραντίνκ. Κακώς δεν ε, προσήθησαν στη δικαιοσύνη, κακώς δεν ήρθαν ε, αντιμέτωποι με τις ευθύνε τους οι υπεύθυνοι. Η αξιοπιστία λοιπόν ε, της, του δικαστικού συστήματος της Τουρκίας από την δίκη αυτή δεν βγήκε αλόβητο και θα πρέπει αυτό να το αναφέρουμε και στην έκθεσή μας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και νομική δικαστική συνέπεια εφόσον υπάρξει μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν τη Ρία για το εξαιρετικό τη έργο και νομίζω ότι από κοινό αύριο θα ψηφίσουμε και θα κρίνουμε μια έκθεση η οποία και θα διαβαστεί πολύ στην Τουρκία και θα είναι και χρήσιμη. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριο uh, Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τη Ρία. Πάρα πολύ δύσκολα και αμφιλεγόμενα όλα αυτά τα θέματα όπως γνωρίζουμε. Αλλά πάρα πολύ καλά τα η Ρία. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πάρα πολύ λεπτά δύσκολα σημεία και το πιο σημαντικό είναι τελικά να σημειωθεί κάποια πρόοδος για τη σχέση μας με την Τουρκία και εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπορούμε να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, αυτό δηλαδή τουλάχιστον να επιτευχθεί πρόοδος είναι υπέρ ημών και υπέρ της Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα τώρα όσοι θέλουν πλήρωζαν να συμμετάσχουν στον δημοκρατικό μετασχηματισμό θα πρέπει να αποκηρύξουν τη βία. Θα πρέπει σε αυτό να είμαστε ξεκάθαροι και συγκεκριμένα ενώ το, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας του ΠΚΚ. Και για την Κύπρο ισχύει αυτό. Θα πρέπει όλοι να κάνουν χειρονομίες, να μην πιέζουμε μόνο την τουρκική πλευρά να προβεί σε παραχωρήσεις όταν δεν υπάρχει αντέλαμο την άλλη πλευρά. Πάντως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιολογητή έκθεση και θα βοηθήσουμε. Ο Χατζηγεωργίου, παρακαλώ. Κύριοι συναδελφοί, να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Νόμου για την δουλειά που έκαμε. Ήμασταν πρόσφατα μερικοί από εμά ω μέλη τη Μιχτή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία στην Τουρκία και υπήρξαμε όλοι μάρτυρε των ε, ε, δεδομένων που έβαλαν μπροστά μα εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων που έκαναν έντονη αναφορά στις ε, φυλακίσεις πέραν των 100 δημοσιογράφων ε, στην Τουρκία, ε, πολλών εκατοντάδων φυλακισμένων εκπροσώπων του κυρδικού κινήματος, με την κατηγορία της επαφής με το KCK που θεωρείται κατά τους ίδιους παρακλάδι του ΠΚΚ, οχτώ βουλευτές της Τουρκίας μέσα στις τουρκικές φυλακές, και μας δόθηκε μια εικόνα τουλάχιστον κατά αυτό το μέρος των συναντήσεων μια Τουρκίας η οποία δυσκολεύεται να βρει τον δρόμο προς την ε, δημοκρατία. Για το κουρδικό ζήτημα ουσιαστικά δεν γίνεται απολύτως τίποτα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι αυτό το θέμα το παρακολουθεί απλώς ε, και δεν πιέζει στο να αναγκαστεί η Τουρκία να λύσει ένα μεγάλο, μεγάλο ζήτημα που αφορά δεκάδες, δέκα και πλέον εκατομμύρια ανθρώπους, 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Τουρκία, επειδή εδώ πολλοί συνάδελφοι έκαναν αναφορά για άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24, και εμεί δεν είμαστε εναντίον τη ενταξιακή διαδικασία τη Τουρκία και του ανοίγματο κεφαλαίων. Θέλω να σα πω το εξή. Εγώ προκάλεσα εκεί τον κύριο Μπαγής να μας πει τι θα κάνει η Τουρκία σε περίπτωση που η Κύπρος κατά την προεδρία της ε, βάλει στο τραπέζι την συζήτηση ανοίγματο κάποιων κεφαλαίων. Θέλω να ενημερώσω το σώμα εδώ, τους συναδέλφους όλους, ότι ο κύριος Μπαγής απήντησε όχι. Δεν ενδιαφέρεται για άνοιγμα κεφαλαίων κατά την διάρκεια της Κυπριακής ε, Προεδρίας. Ουσιαστικά δηλαδή απαγορεύει στον εαυτό της την συνάντηση ή απαγορεύει στον εαυτό της να βρει ένα διάδρομο επικοινωνίας με την Κύπρο. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να καταγγελθεί, να πάει ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν γίνεται απριόρι ε, να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο απέναντι στην Κυπριακή Προεδρία που λέει ότι δεν θα έχει καμιά επαφή μαζί της αλλά απέναντι στο ενδεχόμενο να συζητηθεί αυτό που πολλοί συνάδελφοι βάζουν εδώ πέρα. Η χώρα δηλαδή που καίγεται για άνοιγμα κεφαλαίων ε, συμπεριφέρεται ε, ή απαντά με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να καταλήξω με το εξή. Νομίζω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το δίκαιο μέσα από αυτή την έκθεση και να κληθεί η Τουρκία σταθερά και καθαρά να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο. Δεν έχει να χάσει τίποτε, συνάδελφοι. Δεν έχει να χάσει τίποτε εάν αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο κατά τα ευρωπαϊκά δεδομένα και πρότυπα δεν έχει να χάσει τίποτα. Αλλά είναι υποψήφια χώρα. Επίσης πρέπει να γίνει έντονη αναφορά στην υλοποίηση του ψηφίσματος 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για την παράδοση της πόλης της Αμοχώστου στους κατοίκους της κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με την γραπτή διακήρυξη του Κοινοβουλίου μας η οποία πήρε 50% συν ε, υπογραφές από τους, ε, από τους συναδέλφους. Υπάρχει ένα, μια τροπολογία, αγαπητοί συνάδελφοι, που αναφερόμενη στην αμόχωστο, αναφέρομαι στην τροπολογία 315, παραπλανεί, λέγοντας ότι καλή σε εφαρμογή του 550, δηλαδή της απαστροφής της αμοχώστου, και συμπληρώνει και του Διεθνούς Αεροδρομίου της Λευκοσίας Ερκάν, λέει. Δεν έχει καμιά σχέση, δεν μπορούμε να, να παραπλανούμε για το περιεχόμενο ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Το 550 κάνει μόνον αναφορά στην αμόχωστο. Δεν κάνει καμιά αναφορά σε οτιδήποτε άλλο, χωρί να λέω ότι εμεί δεν μπαίνουμε σε οποιαδήποτε συζήτηση. Κλείνω με τι απειλέ τη Τουρκία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κύπρου. Η Κύπρος έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, η Τουρκία όχι. Και η Τουρκία έχει βγάλει μια ανακοίνωση μόλις προ 15 ημερών του Υπουργείου Εξωτερικών που λέει ότι οι ξένες εταιρείε ε, να μην προσεγγίσουν και να μην διενεργήσουν εξορίξεις στην ΑΟΣ της Κύπρου διότι αυτό θα προκαλέσει την οργή ή την ένταση εκ μέρους της ε, Τουρκίας. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο μας να εκφράσει την πίστη του ότι η Τουρκία μπορεί και πρέπει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες που πρέπει να αναλάβει. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα κατάλογο ομιλητών που μας επιτρέπει να αφιερώσουμε και το απόγευμα σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αφού μίλησαν οι σκιώδεις ηγητές, να περιορίσετε το χρόνο σας σε 1,5 λεπτό, αν συμφωνείτε. Ο κύριος Νταφ θα το αποδείξει ρητά ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, Άντριο, έχεις το λόγο. Well, uh, Mr. President... Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω. Από την, κοινή, από την μεικτή κοινοβουλευτική συνάντηση που είχαμε στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα, θα ήθελα να αντλήσω δύο συμπεράσματα. Πρώτον, οι συνταγματικέ διαδικασίες είναι πλέον πιο πολυφωνικές και πιο προηγμένες από ό,τι εμείς ε, φανταζόμαστε και αυτό θα είναι καθοριστικό για όλα τα υπόλοιπα που θα συμβούν. Και στην Τουρκία την ίδια και στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ε, γείτονες χώρες. Είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε και να εξετάσουμε εντελεχώς και να ενημερωνόμαστε διαρκώς για την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. Ο κ. Τσίτσεκ, ο πρόεδρος της ε, Μεγάλης Εθνοφιανέλευσης που προεδρεύει στην ε, Μεκτή Επιτροπή και είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του κειμένου του συντάγματος, είναι αρκετά θετικός και ευνοϊκά και κείμενο στην ιδέα ότι τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου μπορούν να διαδραματίσουν εδώ κάποιο ρόλο και αυτό είναι καλό και πρέπει να συνεχιστεί. Το δεύτερο σημείο αφορά την Κύπρο. Συμφωνώ ότι η προοπτική του να γίνουν παραχωρήσεις από την Τουρκία προς την Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Οπότε θα πρέπει να να σταθεί εδώ ισχυρή η κυβέρνηση της ε, Κύπρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα πρέπει, νομίζω, και η Κυπριακή, Δημοκρατία του Συμβουλίου, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου να καταγγείλει αυτή την πλόφα των ε, Τούρκων, να τους προκαλέσει. Να δείξει κατά πόσον έχουν ή όχι την προθενία για το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24. Νομίζω αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε αυτή η παραλυσία, η απόλυτη αδράνεια για το κυπριακό ζήτημα να πάψει και να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα τα πω στα Ολλανδικά. Θέλω να ευχαριστήσω τη Ρία καταρχάς και η Ρία όσο κανείς άλλος γνωρίζει ε, πολύ καλά τα πράγματα, ε, καταλαβαίνει πόσο μεγάλη είναι η ελεξάρτηση και είναι κρίσιμη η καιρή και με τη θετική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το επόμενο διάστημα νομίζω θα αποκτήσει και μεγαλύτερη σημασία αυτή η ατζέντα με την Τουρκία γιατί είναι θέμα συνεργασίας. Θα πρέπει ε, από κοινού να συνεργαστούμε. Και η θετική ατζέντα λοιπόν ε, ε, βρήκε ένα σημαντικό χώρο να δώσει στα δικαιώματα των γυναικών. Και εγώ ήμουν την περασμένη εβδομάδα στην Τουρκία και ακριβώς αυτά τα θέματα, θεμελιώδη δικαιώματα, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και γυναικεία δικαιώματα ως υποκεφάλαιο ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό και η ελευθερία της έκφρασης. Αν θέλουμε κάτι να κάνουμε ε, για τον αντιτρομοκρατικό νόμο και τις καταχρήσεις τις οποίες οδηγεί. Θα πρέπει από κοινού με την Τουρκία να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε. Είναι σημαντικά τα κεφάλαια 23 και 24 και είναι σημαντικό πραγματικά να ε, φροντίσουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Έχουμε και εμείς ευθύνη και καθήκον. Και θέλω να εκφράσω και μια ελπίδα θα πρέπει από όλες τις πλευρές να υπάρχει μια προθυμία επίλυσης ε, των πραγμάτων και μπορεί να δοθεί και ένα κίνητρο από την Κυπριακή Προεδρία για να βρεθούν κάποιες ε, λύσεις. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος δεν ανοίγει το μικρόφωνο του. Thank you, President. Ο κ. Μαυρονικόλας. Στο κυπριακό πρόβλημα και θα ήθελα να πω ότι σε αυτήν την περίοδο από την προηγούμενη χρονιά μέχρι σήμερα αυτό το οποίο έχει παρουσιαστεί από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με την προσπάθεια ανεπίλησης του προβλήματος είναι μια έντονη επιθετικότητα η οποία υποδηλώνει και τις βασικές πολιτικές της Τουρκίας των τρόπων αντιμετώπισης της ερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως επίσης και των πρόσφατων αποκλεισμών της Κύπρου σε σχέση με την αμφισβήτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι η κυρία Όμεν έχει πετύχει να παρουσιάσει ένα έγγραφο το οποίο είναι συνενετικό και παράλληλα φαίνεται ότι υπάρχει συνένεση και από όλες τις πολιτικές ομάδες. Έχω την ανάγκη να καλέσω την κυρία Νόουμεν να παρατηρήσει μία πρόταση για τροποποίηση, την 323, η οποία αναφέρεται στον επικισμό. Ο συνεχιζόμενος επικισμός της Κύπρου, που σήμερα αναφέρεται ότι υπάρχουν περίπου 700.000 έπικοι, Τούρκοι έπικοι στα κατεχόμενα, κάθε άλλο παρά διαμορφώνει καλό κλίμα για τη λύση του κυπριακού προβλήματος εάν συνεχίσει αυτή η δημογραφική αλλαγή της Κύπρου δεν θα υπάρξει τρόπος να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα. Γι' αυτό προτείνω στην κυρία Νόουμεν έναν amendment το οποίο έγινε αποδεκτόν και στα προηγούμενα δύο χρόνια που καλεί την Τουρκία να σταματήσει των παράνομων επικισμών των κατεχομένων. Αυτή είναι μια επιθετική πολιτική η οποία οδηγεί στην τουρκοποίηση της Κύπρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη και να μην επαναλάβω τους επένους προς την εισηγήτρια. Αν σας πω τα εξής πρώτα. Πρώτα όσον αφορά το κουρδικό. Κυρία Ομιν Ράιτον Στην παράγραφο 22 τα βλέπει πάρα πολύ ζυγισμένα τα πράγματα. Τα ζύγισε καλά εκεί που λέει για την ε, αναγνώριση και την πολιτική λύση στο κορδικό. Όμως θα πρέπει να ξανακοιτάξει την παράγραφο 33 όσον αφορά την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι, εδώ πέρα είπαμε ότι έχουμε μια σειρά τροπολογιών από τους φιλελευθέρους και από άλλους 34 με 38. Παρακαλώ, ε, ρίξτε μια ματιά. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες συλλήψεων κατά χρόνο του νόμου. Ε, κύριε Φανούρτη, και αναφερθήκατε σε αυτό. Τελικά δεν υπάρχει κανένας πολιτικός χώρος, ε, ούτως ώστε να υπάρχει κάποιο είδους ε, νόμιμη εκλογή πολιτικού Κούρδου, ο οποίος να μπορεί να ανέβει στην πολιτική σκηνή. χρησιμοποιείται μέσα στην τρομοκρατική νομοθεσία και κατά αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε σε μια πολιτική λύση. Δεύτερον, για την Κύπρο. Δεν συμφωνώ ότι εδώ πέρα τα λέει καλά η κυρία Όμεθ, χρειάζεται να αλλάξουμε την παραγραφό 25 συγκεκριμένα. Τουλάχιστον να αναγνωριστεί η αθετημένη υπόσχεση του 2004 που είχαν υποσχεθεί ελεύθερο εμπόριο και να σταματήσει η απομόνωση του τουρκικού τομέα. Και συμφωνώ με τα όσα είπε ο Άντριου Ντάφ για την Κύπρο επίση. Μεγάλη μου χαρά. Η, κυρία Μενερό ήταν εδώ. Είπε ότι θα λάβει υπόψη την τροπολογία για το 34, ούτω ώστε να ξαναγυρίσουμε πάλι σε ε, ε ελεύθερο καθεστώ όσο αφορά τι θεωρίε διαβατήρια. και επίσης και τα δικαιώματα ομοφυλοφίλων ε, και λοιπά για το 24. Σω. Σας παρακαλώ λίγο μεγαλύτερη πειθαρχία χρονική, αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε και τη Σερβία μετά. Ο κύριος Πέτρελε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τα συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια. Νομίζω ποτέ δεν είχαμε τόσο συγκεκριμένη έκθεση, με τέτοια ακρίβεια, ε, που να περιγράφει τόσο ε, κριτικά την κατάσταση, αρχής γενομένης από την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης. Η έκθεση είναι τις πρόοδους που έχουν γίνει, αλλά και έκθεση που πρέπει να γίνει. Πολύ σημαντική είναι η υποστήριξη της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος, θα πρέπει να ανοίξει το κεφάλαιο για τη δικαιοσύνη και το θέμα της ε, ε, ελεύθερης ε, κυκλοφορίας χωρίς θεώρηση διαβατηρίων για ένα χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ συγκεκριμένα στοιχεία αυτά. Επιτρέψτε μου να κάνω και μερικά γενικά σχόλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Τουρκία να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος με δημόσιο διάλογο, μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος επίσης. Τους τελευταίους μήνες η ε, αντιπολίτευση είναι σε πολύ πιο στενή επαφή με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τώρα επειδή επίκυνται διάφορες εκλογές, ε, θα ήταν χρήσιμο εκατέρωθεν να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, αλλιώς ε, στη συνέχεια μπορεί να επιβραδυνθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Νομίζω ότι προσπάθησε να δώσει κάποια στοιχεία πιστικά και εξισορροπημένα για πρώτη φορά. Βλέπουμε το Συμβούλιο το οποίο καλείται να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να ξεκινήσει ο διάλογος για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων διαβατηρίων. Είναι η μόνη χώρα που πρέπει να παίρνουν οι κατοικοί τη θεώρηση, ενώ είναι συνδεδεμένοι, ε, είναι σε προενταξιακό καθεστώς. Είναι απαράδεκτο αυτό όσον αφορά την επαφή του κόσμου, να έχουμε μια υποψηφία χώρα η οποία τις οποίες οι κάτοικοι μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα. Έλαβε υπόψη αυτά που είπε ο κ. Νταφ και η Λέδη Λάτφορτ ε, είπαν ότι είναι εξορροπημένα τα πράγματα. Εγώ δεν συμφωνώ. Νομίζω θα πρέπει περισσότερο να λάβουμε υπόψη ε, τι υποσχέσει ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τη στηρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτέ τι υποσχέσει που έδωσε τον Απρίλιο 2004 και έτσι να σταματήσει η απομόνωση τη τουρκοκυπριακή κοινότητα. και να δοθεί μια συνολική λύση. Μια λύση πριν την αρχή της Κυπριακής Προεδρίας. Πώς θα υπάρχει Προεδρία χωρίς να μπορούν να συμμετάσχουν εκεί οι Τουρκοκύπροι. Δεν έχει νόημα. Κύριος Ρότσεκ. Já bych chtěl též pogratulovat zpravodajce za velmi vyváženou. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για το ότι είναι αντικειμενική αυτή η έκθεση, είναι εξισορροπημένη, είναι θετική και εδώ πέρα αναγνωρίζεται η πρόοδο που έχει σημειωθεί από πλευρά τη Τουρκία. Ήταν βήμα πρόοδο οι εκλογέ που έγιναν πέρσι και αναφέρονται εδώ πέρα το ότι υπάρχουν ευκαιρίε, υπάρχουν δυνατότητε τώρα, ούτω ώστε να καταλήξει η Τουρκία στο να έχει ένα νέο σύνταγμα. Επίση, έχουμε και το θέμα τη ε, τουρκική δικαιοσύνη. Εδώ υπάρχουν κάποιε επικρίσει όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Τώρα, συγκεκριμένα, θα ήθελα να σα αναφέρω κάτι για το Κυπριακό. Νομίζω ότι η έκθεση. Επ' αυτού επίσης τα λέει πάρα πολύ εξισορροπημένα ε, νομίζω ότι λαμβάνει υπόψη τα επιχειρήματα των μεν αλλά και των δε. Η Τουρκία. Εάν δεν μπορεί να συνομιλήσει με την Προεδρία της Προεδρίας, δηλαδή την Κυπριακή, τότε καταλήγει σε αντιπαραγωγικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να μπορεί να κάτσει στο τραπέζι, θα πρέπει να προχωρήσουν οι σχέσει με την Κύπρο. Φυσικά και σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, αναφέρεται εδώ πέρα η έκθεση στην στρατηγική σημασία τη χώρα. Ορθώ εδώ καλείται η Τουρκία να ανοίξει διάλογο με Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Επίση καλείται η Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο και να μπορεί να συμμετάσχει στην άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Ε, αναφέρεται επίση και το Μεσανατολικό. Έχουμε ζητήματα εδώ και με τα Δυτικά Βαλκάνια, Πακιστάν, Ιράν. Θα πρέπει για όλα αυτά τα ζητήματα να υπάρχει στενή συνεργασία Τουρκία-Ένωση. δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, στην πρόοδο σε αυτά τα μέτωπα το κυπριακό. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, όλοι να έχουν μια επικοδομητική στάση, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει και τις δύο κοινότητες. Αλλά και ο ΙΕ θα πρέπει να βοηθήσει να ολοκληρωθούν οι σχετικές συνομιλίες. Ευχαριστώ. 78% ήταν υπέρβαση του χρόνου σας. Κοιτάξτε αγαπητοί συνάδελφοι. Κάπως πρέπει να το συμμαζέψουμε. Δεν θα προκάνουμε. Δεν μ' αρέσει να σας κόβω το μικρόφωνο, αλλά σας παρακαλώ κοιτάξτε λίγο το χρόνο σας και φροντίστε. Ο κύριος Κουμουτσάκος παρακαλώ. Thank you, Chair. Um, I Ευχαριστώ Πρόεδρε να συγχαρητηριά για το εξαιρετικό της έργο που συντάσσει πάλι μια πολύ καλή ισορροπημένη έκθεση για άλλη μια φορά φέτο και ήθελα εδώ να παρατηρήσω το εξή. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Οι δαπάνες του 3,5-4% του ΑΕΠ ε, ε, δαπάνε ε, για τον αμυντικό εξοπλισμό, στον οποίο έχει ξαναγκαστεί η Ελλάδα εδώ και δεκαετίε, είναι ένα από του λόγου για τι πολύ δυσχερεί οικονομικέ συνθήκε που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Είναι σαφέ, συνάδελφοι, ότι η Ελλάδα δεν πάσχει από εθνικό μαζοχισμό. Δεν μα αρέσει να ταπανούμε δι επί δι ευρώ για αμυντικό εξοπλισμό. Η Ελλάδα πιστεύει και έχει κάθε λόγο να θεωρεί ότι αντιμετωπίζει μια πραγματική και διαρκή απειλή εξ Αυτά είναι τα λόγια του ίδιου του Υπουργού Άμυνάς μας. Επιπλέον, η Τουρκία με την πολιτική της διαρκών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου και της παραβίασης ε, της θαλάσσιας, ε, των θαλάσσιων και ενέριων σύνορων του Αιγαίου επαναλαμβάνει αυτές τις απειλές και τις κάνει να διαρκούν. Γι' αυτό λοιπόν, συνάδελφοι, και για τις πρόσφατες απειλές κατά της, δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις εντάσεις, την κλιμάκωση των εντάσεων με το Ισραήλ, τη Συρία και το Ιράκ, σημαίνει ότι η στρατιωτικοποίηση έχει γίνει ένα απόσπαστο στοιχείο της πολιτικής ε, εξωτερικών υποθέσεων της Τουρκίας. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να γνώμουμε αυτή την κατάσταση πρέπει να αποσταλεί ένα σαφέ μήνυμα και προ τον ελληνικό λαό, που αυτή τη στιγμή των τεράστιων θυσιών που καταβάλουν, το Ευρωκοινοβούλιο τουλάχιστον, αποθαρρύνει και μάλιστα αποθαρρύνει έντονα την Τουρκία, αποδοκιμάζει μάλλον την Τουρκία για τις διαρκείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του ενέργειου χώρου του Αιγαίου. Δεν μπορεί η Ελλάδα να εξαναγκάζεται να εξακολουθεί αυτέ τι βάσταχτε αμυντικέ δαπάνε σε ένα τόσο δυσκερέ οικονομικό περιβάλλον. Ευχαριστούμε, ο κ. Παπαδόπουλο. Μίση. Κυρία Παπαδόπουλο, αντίγωνα. Κύριε Πρόεδρε, λυπούμε γιατί μιλούμε ότι η Κύπρος είναι πρόβλημα για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας δεν υπάρχει πρόβλημα για την ενταξιακή πορεία της τουρκίας αν η ίδια η τουρκία αντιληφθεί ότι στην περίπτωση της κύπρου είναι ο θήτης. η κύπρος η χώρα μου είναι το θύμα. είναι θύμα μιας τουρκικής εισβολής του 1974 που συνεχίζεται για 38 χρόνια. η τουρκία στην περίπτωση της κύπρου απειλεί την κύπρο να μην εξορίξει πετρέλαιο στη δική της ΑΟΣ. συνεχίζει τον παράνομο επικισμό. εξακολουθεί να ε, να καταπιέζει ανθρώπινα δικαιώματα προσφύγων και αγνωμένων. Και δυστυχώς όταν μιλούμε για το Κυπριακό η Τουρκία είναι η δυνατή χώρα και θα έπρεπε οι εκκλήσει μας να είναι η ίδια η Τουρκία να σεβαστεί το πρωτόκολλο της Άγκυρας, να το υλοποιήσει, να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να μην εκτοξεύει οι άπειλες. Εμείς θέλουμε να ανοίξουν τα κεφάλια. Για να ανοίξουν κεφάλια όμως πρέπει να σεβαστούμε ότι υπάρχει μια διακυβερνητική ε, διαβούλευση και χρειάζεται το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Το μικρόφωνο, το μικρόφωνο σας. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλάν μόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ να συγχαρώ όπως οι άλλοι συνάδελφοι την ε, Ρία για ε, το ραντεβού τέλεσε. Βέβαια έχουμε όλες αυτές τις 500 περίπου τροπολογίες. Τέλος πάντων, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και απλώς θα ήθελα να σας πω μια παρατήρηση και θα ήθελα κάτι να ζητήσω, μια διευκρίνηση. Η παρατήρηση μου είναι η εξής. Ε, θέλω να σας πω κάτι για τον συμβασμό 23 ε, όσον αφορά ε, τις βίζες των διαβατηρίων. Ακριβώς ε, όπως τα είπαμε, έχουμε και το θέμα του mail που τα είπαμε μέρα ότι θα πρέπει να το πώς να τον έχουμε μια σύγκληση των πολιτικών. αυτή η σύγκληση που τη ζητάμε είναι πάρα πολύ αμφίσιμη, πάρα πολύ αμφισβητούμενη. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη χώρα που είναι χώρα υποψήφια. Χρειάζεται να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Τα, τα, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, δεν ξέρω αν μου το επαληθεύσετε, αλλά διάβασα ότι ο, ε, Συρία, Λιβύη, ε, Σουδάν, Πακιστάν είναι χώρες ε, στις οποίες έχει άρει το καθεστώς, τη ρύθμιση που είχε πριν το Ιατροφείο Υπουργείο των Εξωτερικών. Επομένω, θα πρέπει να, να γίνει ε, πιο ξεκάθαρη αυτή η τροπολογία. Στο 14 υπάρχει εδώ πέρα μία παράγραφος που λέει κάτι λέει για διατάραξη της ειρήνης κλπ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν ξέρω απ' έξω τι τη τα των δικαιώματα, αλλά εδώ πέρα με, με εκπλήσει αυτή η παραπομπή. Με εκπλήσει αυτό το οποίο εδώ πέρα διατυπώνεται. Κύριε Χάουιτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια. Μου έστειλε ένα πάρα πολύ μεγάλο mail χθε. Θα το μελετήσω και θα τη απαντήσω. Άκουσα και το... Θέλω επίση να σα πω κάτι για εκ μέρου του κ. Μπιόλ, ο οποίο απουσιάζει. Ναι. Έχω υποβάλει κάποιε τροπολογίε. Τόσο, κάποιες από αυτές θα είναι προσθήκη, θα επανεχωρηθά. Επίσης, όσον αφορά τους αντιρρησίες συνείδησης, έχουμε κάποιες παρατηρήσεις και όσον αφορά επίσης τα συνδικάτα. Στο 22 τώρα. Συμφωνώ με τα όσα ελέγχθησαν και όσον αφορά το KCK έχουμε κάποιες συλλήψεις, κάποιες παραπομπές ε, και αυτές οι λεγόμενες προφυλακίσεις κρατάνε πάρα πάρα πολύ. Έχω μια σχετική τροπολογία. Και τώρα ο 97 επίσης, ξανακοιτάξτε τη συμβαστική διάταξη. Νομίζω ότι εδώ είμαστε ε, συνεπείς με αυτό που είπε ο κύριος Φανόρνταν, αλλά και ο κύριος Λάμστροφ σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ πρέπει να είμαστε κάθετοι κατηγορηματική. 24 επίσης για την εξωτερική πολιτική, το 25. Δεν ζητούμε εδώ απλώς νομοθεσία. Η εφαρμογή των όσων για τα βασανιστήρια. Απλώς θα πρέπει όμως εδώ πέρα να ληφθεί υπόψη τροπολογία μου ή να μπει ως προσθήκη. Ευχαριστώ. Κράσιλερ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή μπορεί να συνεισφέρει να λύσουμε το γόρδιο δεσμό μεταξύ Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών της Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Αλλά υπάρχει και η αρχή του δούνε και «Δεν ε, Σου δίνω κάτι, μου δίνεις κάτι. Μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του 2004. Πώς δεν ανταποκρίθηκε. Κοιτάξτε, και το πρωτόκολλο της Άγκυρας ακόμα δεν υλοποιείται. Συνεχίζεται ο παράνομος επικισμός. Εμένα μου θυμίζει τον παράνομο επικισμό του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Ισχύει αυτή η σύγκριση. Δημιουργούνται τελεσμένα που δεν μπορούμε έτσι να τα εγκρίνουμε. Και εγώ Συμφωνώ να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά ε, πρέπει σε αντάλλαγμα να δοθεί κάτι και μάλιστα ταυτόχρονα. Να βγούμε από αυτό το δίλημα ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση. Και αν δούμε τι δηλώνει η σημερινή τουρκική κυβέρνηση, ελπίζω λίγο να μετριαστούν οι δηλώσεις αυτές, γιατί δεν μπορεί ένα κράτος μέλος να αναγνωρίζεται, να λέει μια χώρα ότι εγώ θέλω να μπω στην Ένωση αλλά με την τάδε χώρα μέλος δεν διαπραγματεύομαι. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Εγώ ανέκαθεν ήμουν υπέρ της ένταξης της Τουρκίας, θα εξακολουθώ να το πιστεύω, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια ισοτιμία στη δράση. Όλα τα άλλα θετικά αρνητικά τα είπε θαυμάσια η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Κάτσιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι θεωρώ πολύ σημαντικό τα μέλη του ε, τουρκικού κοινοβουλίου να έρχονται εδώ στις ε, Βρυξέλλες ε, συστηματική βάση, διότι είναι σημαντικό να παρατηρούν τι γίνεται εδώ. Ε, όλο και περισσότεροι επισκέπτε έρχονται και από την Άγκυρα επίση και αυτό δημιουργεί μια πολύ καλή ατμόσφαιρα για το μέλλον. Θέλουν να παραδειγματιστούν. Ε, θέλω απλώ να επισημάνω το γεγονό ότι τον Ιούλιο θα ανοίξουν δύο κεφάλαια για την περίπτωση του Μαυροβουνίου, του 23 και 24. Αυτή είναι η νέα προσέγγιση και στρατηγική μα. Η νέα στρατηγική απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κάποιο τρόπο. Εάν ισχύσει κάτι και για τη Μακεδονία, θα πρέπει κάτι ανάλογο να γίνει και για τις υπόλοιπε υποψήφιες χώρες για όσους διαπραγματεύονται ή πρόκειται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να αρχίσουμε επιτέλους με το κεφάλαιο 23 και 24. Το κεφάλαιο 23 θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα ευαισθητότερα προβλήματα και νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτελέσουμε πρόοδο στην περίπτωση της Τουρκίας και στη σχέση μας με τη χώρα αυτή και να έχουμε μια πολύ καλύτερη ατμόσφαιρα όχι μόνο στην ίδια τη χώρα αλλά και στην περίπτωση της Κύπρου. Εδώ αφορά αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα μέσα μαζική ενημέρωση, την κατάσταση στις φυλακές, την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, ό,τι για μας είναι ζωτική σημασία προκειμένου να υπάρξει ένταξη, η πορεία ένταξης και τελική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόοδος όμως απαιτείται. Και τα κεφάλαια 23 και 24 είναι οι μαγικές λέξεις, πιστεύω εδώ. Thank you very much. Now, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Φιλόρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Yes, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Συγγήτρια, μέλη της Επιτροπής, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέψτε μου να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια για την ε, πολύ ε, ισόρροπη έκθεση που έχει συντάξει ως τώρα νομίζουμε ότι απεχεί πολύ σωστά και τη δική μας την αποτίμηση στην ε, τελευταία, την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση πρόοδου. Εάν μου επιτρέπετε Πρόεδρε, θα ήθελα να περιοριστώ στις τροπολογίες όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται ρητός. Καταλαβαίνω ότι η συμβαστική πρόταση 5 περιέχει την ε, αίτημα να ξαναδούμε στην επόμενη έκθεση του 2012 τις τροπολογίες, τις συνταγματικές τροπολογίες που έγιναν το 2010. Βεβαίως και πρόκειται να παρακολουθήσουμε τη συμμόρφωση της Τουρκίας με τα πολιτικά κριτήρια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται σεβαστά. Έπειτα, στην συμβιβαστική τροπολογία 11 όπου ζητάτε συγκεκριμένο παράρτημα και λεπτομερή ε, πορίσματα για την περίπτωση εργένεκων. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να ελέγχει την λειτουργία του δικαστικού συστήματος υπό το φως των ανάλογων αρχών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια και την δίκαιη μεταχείριση από το δικαστικό σύστημα. Εδώ η Επιτροπή δεν μπορεί να δει τις λεπτομέρειες υποθέσεων όπως η Εργένεκον, αλλά μόνο ζητήματα ισότητα ή αδικίας, παρανομίας. Εδώ αυτά θα περιλαμβάνονται στα πορίσματα της ε, μελλοντική μας ε, της έκθεσης πρόοδου και της έκθεσης ε, για την Τουρκία που θα είναι έτοιμη το φθινόπωρο. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και οι λεγόμενες peer reviews, οι εκθέσεις όπως αυτή που ήδη ετοιμαστήκε για το 2011 στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Τουρκία και ευχαρίστως να σας την ε, μεταδώσω το η δεύτερη έκθεση αυτού του τύπου για το πώς λειτουργεί το δικαστικό σύστημα και τα δικαστήρια για σοβαρά αδικήματα που ασχολούνται με σοβαρές υποθέσεις όπως η Εργένα, η Κόνης, Χάμερ και ούτω καθεξής. Αυτή η έκθεση ήδη έχει αρχίσει να ετοιμάζεται και πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σπότμαν από το ιδιαίτερο γραφείο της ΥΠΑΤΗΣ εκπροσώπου που ε, ε, είναι επιφορτισμένος με θέματα εξωτερικής πολιτικής και συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να καλωσορίσω το έργο της εισηγήτριας και να πω πόσο Ικανοποιημένοι είμαστε, ιδίω με την παράγραφο 36 που αναφέρεται στο στρατηγικό ρόλο τη Τουρκία και τι δυνατότητε ε, σχέσεων συνεργασία μέσω τη εξωτερική πολιτική τη χώρα αυτή. Η Τουρκία παραμένει μια βασική προτεραιότητα για την υπατή πρόσωπο και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως με τις σχέσεις μας με την Τουρκία λόγω της Αραβικής Άνοιξης αλλά και επειδή είναι ένας σημαντικός φορέας για να αναπτύξουμε το διάλογο εξωτερικής πολιτικής μας και έναν θετικό κατάλογο προτεραιοτήτων. Νομίζουμε ότι, θεωρούμε μάλλον ότι το έργο του Κοινοβουλίου ενθαρρύνει πραγματικά και τονώνει τι προσπάθειε για την για να υπάρχει σύμπλευση τη ε, εξωτερική πολιτική τη Τουρκία με αυτήν τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, υπάρχει θετική μνήμα στην έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Όμεν Ρόιτεν. Έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αρχίσω από το τελευταίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτικής Δράσης για τα καλά τους λόγια. Όσο γίνεται ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε καλή τη συνεργασία μας. Στη συνέχεια, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνομαι. Κάντε λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Στον κύριο Φιλόρη, κατανοώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και κάποια παλιά αντανακλαστικά. Τη στιγμή που το Κοινοβούλιο ζητάει να μας δώσετε λεπτομέρειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντάει ότι δεν είναι δωρεάν αυτή η παροχή. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Όταν ρωτάω κάτι θέλω να μου απαντούν. Τι σημαίνει αυτή η απάντηση. Ε, το Κοινοβούλιο έχει απορίες, θα πρέπει να τις απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι για την παρατήρησή σας ότι είναι η έκθεση καλή και ισόρροπη. Τα βασικά σημεία των ε, συναδέλφων πρόεδρε ποια ήταν. Πρώτον, η Τουρκία θα πρέπει να διατηρεί καλές σχέσεις με τους γείτονές της. Το είπα και από την αρχή. Αυτό που γράφει για την Κύπρο και εν ώψη της μελλοντικής Κυπριακής Προεδρίας είναι ένα μήνυμα ε, πρακτικό και σαφές. Με μία εξαίρεση, το κύριο ε, Χατζηγεωργίου, ε, πιστεύω ότι άλλοι το υποστηρίζουν. Κύριε Χατζηγεωργίου, κάνετε κάποιες παρατηρήσεις. Κοιτάξτε την παράγραφο ξανά, παρακαλώ. Γιατί ακριβώς και στο πρώτο σχέδιο το είχαμε συζητήσει και ε, το θέμα και με την Κυπριακή Προεδρία την επόμενη και για τους ε, ε, αγνοουμένους αναφέρομαι και στην αμόχωστο. Αυτά που λέτε εγώ τα έχω συμπεριλάβει. Γιατί τα επαναλαμβάνετε. Στη συνέχεια δεν θα πρέπει να παραγνωρούμε και να παραγνωρίζουμε, και το λέω και στη Βαρόνη Λάτφορτ και σε άλλους, ότι υπάρχουν ευαισθησίες, εκατέρωθεν. Και θα πρέπει να ε, δούμε τι λένε οι δύο πλευρές. Η μία λέει ότι σωστά ε, η ε, Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να την προστατεύουμε και η άλλη πλευρά λέει για μια στιγμή τι θα γίνει με την Τουρκία. Και εγώ ως εισηγήτρια οφείλω αντικειμενικά να περιγράφω την κατάσταση. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι δύο όψεις του νομίσματος και δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Και έρχονται πολλές τροπολογίες. Και έρχονται ε, πολλές τροπολογίες που εντάσσονται στην κατηγορία Κύπρος αλλά δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Είπαμε, η έκθεση είναι και αντικειμενική και ισόρροπη. Ε, αυτά τα λόγια κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν. Μετά. Κάτι που με στεναχώρησε λίγο ήταν οι παρατηρήσεις του φίλου μου Φρανσίσκο Μιλάν Μον που λέγει ότι ε, και έχει δίκιο βέβαια η Τουρκία έχει κάνει κάποιες συμφωνίες θεώρησης διαβατηρίου με τρίτες χώρες. Και τη στιγμή που η Τουρκία δεν το κάνει σε διάλογο και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι πρόβλημα. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά υπάρχει και εδώ η άλλη όψη του νομίσματος και η άλλη όψη λέει ότι έχουμε μια έκθεση και λέμε ότι τη στιγμή που η επανεισδοχή έχει υπογραφεί ως συμφωνία μπορούμε να απελευθερώσουμε τις θεωρήσεις διαβατηρίων ή, εν να το δρομολογήσουμε ε, προς τα εκεί και να το συνεννοηθούμε. Ε, μερικοί δυσκολεύονται να το προωθήσουν αυτό. Και πάλι είναι το θέμα της λεπτής ισορροπίας που θα πρέπει να βρω. Μπορώ να απαιτήσω εγώ από κάποιον να κάνει τα πάντα ευθυγραμμιζόμενος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά όταν πρέπει εγώ να κάνω κάτι, δεν κάνω αυτό το βήμα προς την απελευθέρωση της θεώρησης. Καταλαβαίνεις, κάθε φορά είμαστε σε αυτή τη λεπτή ισορροπία. Ζητώ συγγνώμη για τη διατύπωση, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τα διάφορα μελήματα και τις ανησυχίες των πλευρών. Άλλο θέμα. Η έκθεση επικεντρώνεται σε αυτό που είπαν εδώ οι συνάδελφοι, δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, από τα σημαντικότερα ε, κριτήρια της Κοπενχάγης, κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του προσώπου, του ατόμου, αλλά και των συλλογικών κοινοτήτων. Αυτή είναι η καρδιά της ευρωπαϊκής συνεργασίας και θα πρέπει να παραμείνει η καρδιά των μεταρρυθμίσεων που οφείλει να κάνει η Τουρκία. Και στην έκθεση αυτή το τονίζω πάρα πολύ έντονα. Αλλά Τη στιγμή που το κάνεις αυτό και ζητάς από την Τουρκία να κάνει τις μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθούν τα πράγματα και να κατοχυρωθούν καλύτερα στην εθνική νομοθεσία, τη στιγμή λοιπόν που το ζητάς αυτό και στέλνει έκθεση η Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι καν σε θέση να την αξιολογήσει ε, κάπου χωλαίνει η κατάσταση. Δηλαδή, και στα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν του ζητούμε να κάνουν κάτι, θα πρέπει να φροντίσουμε να το επαληθεύουμε και να κοιτάμε ποια είναι η προθυμία και για τα κεφάλαια 23 και 24. Αυτό, αυτό λέμε. Και πάλι νομίζω ότι είναι ισόρροπη η διατύπωσή μας. Συμφωνεί η συγκήτρια με όλα αυτά ε, που είναι τώρα στους, συμβια... συμβιβασμούς, συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν κάποιος είναι εισηγητής, παραμένει μέλος πολιτικής ομάδας. Αλλά θα πρέπει να φροντίζει και ο εισηγητής να επιχείται και να αντανακλάται η θέση του Κοινοβουλίου κατά πλειοψηφία. Για να σταλεί ένα μήνυμα ε, στους ανθρώπους με τους οποίους διαπραγματευόμαστε θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα σαφές, δυναμικό, αντικειμενικό, ισχυρό, να εντοπίζει τα στρεβλά του συστήματος, να τα κατονομάζει, αλλά ταυτόχρονα να φροντίζει αυτά που πρέπει να βελτιωθούν και βελτιώνονται, να τα αναφέρει. Προσπάθησε η συγκήτριά σας να το πράξει και είμαι ικανοποιημένη που σε γενικές γραμμές νομίζω ότι τα κατάφερα και με υποστήριξαν οι συνάδελφοι κατάλογο ψηφοφορία για αύριο νομίζω είναι θετικό και θέλω να πω και σε κάποιου συνάδελφου. αν μου ζητάτε να αλλάξω κάτι ε, για την ψηφοφορία και το λέω στον Βρετανό συνάδελφο δεν γίνεται αυτό γιατί έχουμε κάνει συμβιβασμούς, ε, κουραστήκαμε πολύ και αν κάποιο δεν θεωρεί ότι η τροπολογία του έχει συμπεριληφθεί καλά σε μια συμβαστική, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορώ 100% να ικανοποιώ του πάντε. Αλλιώς δεν θα μπορούσα ποτέ να συντάξω έκθεση για την Τουρκία. Ευχαριστώ. for a very short intervention, please. Very short. I'm Για μια πολύ σύντομη παρέμβαση, κυρία Λάντφορντ. Ε, με συγχωρείτε, πολύ σύντομα, αλλά νομίζω ότι υπήρξε παρανόηση για το τι συμβαίνει με τι θεωρήσει. Εάν η απελευθέρωση των θεωρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Τουρκία ισχύει, αυτό ε, θα πει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζεται να έχουν θεώρηση για να ταξιδεύουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρχει βέβαια έλεγχο διαπατηρίων στα εξωτερικά σύνορα, όμω σε καμία περίπτωση δεν θα ε, κάλυπτε αυτά τα ταξίδια μέσω Τουρκίας. Όποιος δεν είναι Τούρκος υπήκος και ταξιδεύει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέσω Τουρκίας δεν θα καλύπτεται. Αυτό για να καθησυχάσουμε το φόβο ότι δεν θα εξαιρούνται όλοι όσοι περνάνε από την Τουρκία από την υποχρέωση να έχουν θεώρηση. Όχι. Αυτό απηχεί και μια από τις μέρημνες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Δεν θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση για όλους. Όσοι δεν χρειάστηκαν θεώρηση για να περάσουν, ε, να φτάσουν μάλλον στην Τουρκία, δεν σημαίνει ότι απελευθερώνονται από την υποχρέωση να έχουν θεώρηση. Λοιπόν, να μην ανοίξουμε τώρα καινούργια συζήτηση. Σας παρακαλώ, τα είπαμε αυτά, κύριε Χάουτ. Διαδικαστικό, καμία σχέση με το προηγούμενο. Δέχομαι πλήρω ότι η κυρία Όμερόιτ θα πρέπει να γνωρίσει κάποια πράγματα και να δεχτεί κάποια άλλα για να περάσει σε συμβιβασμού. Θυμάστε πέρσι, είχαμε τεράστιο πρόβλημα στην ψηφοφορία, γιατί είχαμε ακούσει ότι ορισμένα πράγματα καλύπτονται από τι συμβιβαστικέ και δεν καλύπτονταν. Παρακαλώ λοιπόν ε, να το κοιτάξει η Γραμματεία, να ε, το φροντίσει στον κατάλογο ψηφοφορία. Εάν δεν αναφέρεται μια διατύπωση, δεν καλύπτεται συμβαστική, να βεβαιωθείτε ότι όλα θα γίνουν εντάξει. Ναι, αλλά χτε το διαπραγματεύτηκα αυτό, λέει η Ριόμεν, με τον κύριο Ραμόνο Μπιόλ και ελπίσαμε και ο κύριο Χάουιτ που ήρθε αργότερα και δεν άκουσε αυτά που είπε η κυρία Γκόμε να τα ε, υιοθετεί. Να το δουν μεταξύ τους παρακαλώ. Εντάξει, θα περιμένω να είναι εδώ και η κυρία Γκόμες, λοιπόν, για να συνεννοηθούμε. Ε, Um, Ευχαριστώ συνάδελφες. Προχωρήσουμε τώρα στην έκθεση για τη Σερβία. Ο πρώτος που έλαβε το λόγο είναι ο εισηγητής. Αφού φύγουν όσοι δεν ενδιαφέρονται από την αίθουσα. Not all of them, not all of them. On Serbia. On Serbia, okay. Okay. Okay. Please, colleagues, let's move on. Not out. Συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε. Όχι εκτός αίθουσας, αλλά στο επόμενο σημείο. No, no, no, no, not yet, not yet. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δεν είναι όριμη η κατάσταση. Συνάδελφοι, παρακαλώ όσοι θέλουν να συζητήσουν, εκτός αίθουσας παρακαλώ, όσοι θέλετε να παραμείνετε, ε, επιτρέψτε μας να εργαστούμε. Επιτρέψτε μας να έχουμε κάποια ησυχία. Χρειάζεται περισσότερο κύρος. I think you have Ε, you have the floor. Κύριε Κάτσιν, το λόγο. Πρόεδρε ε, Πάσκου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τα μέλη της Γραμματείας ε, της Επιτροπής μας ε, και την Εύα Μαρ που εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά Θέλω να ευχαριστήσω και τους βοηθούς και συνεργάτες μου, το γραφείο μου και τους κοιόδες ηγητές, γιατί ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και καλή η συνεργασία και ευρεία η συνένεση για το τελικό ψήφισμα. Με μεγάλη ικανοποίηση και περηφάνεια μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη ατμόσφαιρα να συζητούμε σήμερα για τη Σερβία. Έχει κάνει μεγάλες πρόοδους σε σχέση με προηγούμενους μήνες βάσει τριών κριτηρίων που είναι προϋποθέσεις για την ένταξη μιας χώρας. Συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και ε, συνιστά να δοθεί καθεστώς ε, υποψήφιας χώρας στη Σερβία ακριβώ γιατί έκανε μεγάλες πρόοδους. Συμφωνία για περιφερειακή συνεργασία με την Πρίστινα ε, προχωρεί καλά, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή του τεχνικού πρωτοκόλου για την εφαρμογή των συμφωνιών για την κοινή διαχείριση συνόρων. Ε, ε, συνεργασία με την K4 και τη Ulex επίσης προχωρεί, έχουν φύγει τα οδοφράγματα από τη σερβική πλευρά και έχουν ε, αρχίσει διώξει ε, για του υπεύθυνου των επεισοδίων του περασμένου Ιουλίου. Αυτό δείχνει την προθυμία του Βελιγραδίου να εξομαλύνει τη σχέση του με την Πρίστινα. Αυτό θα πρέπει να το πούμε και να το τονίσουμε και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει καθεστώς ε, υποψήφιας χώρας στη Σερβία. Λυπάμαι που ορισμένα κράτη-μέλη τελευταία στιγμή προσπαθούν να μπλοκάρουν αυτό το θέμα. Ε, γιατί είναι κρίμα τελευταία στιγμή και με τέτοιο τρόπο. Η έκθεση συμπληρώθηκε από τροπολογίες και προφορικές και παρακαλώ τους συναδέλφους ε, αύριο να μην καταψηφίσετε τις προφορικές τροπολογίες, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κείμενο ε, πολιτικά εύστοχο. Επιτέλους η Σερβία παίρνει τον δρόμο της ευρωπαϊκής ένταξης και θέλουμε να επικεντρωθούμε ε, στο κράτος δικαίου, στην καταπολέμηση της συστημικής διαφθοράς. Επί σειρά ετών οι μεταρρυθμίσεις ε, καθυστερούσαν στη Σερβία λόγω πολιτικής εμπλοκής και του κοσυφοπεδίου και υπήρχαν επίσης δυσκολίες στη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η κατηγορούμενη σήμερα είναι ενώπιον του δικαστηρίου και μπορεί να συμμετέχει η Σερβία στη διεθνή κοινότητα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ε, προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικοί ηγέτες δεν θα έχουν πλέον δικαιολογία για να μην εξυγχρονίσουν τη χώρα. Είναι πολλές ε, υποθέσεις στη δικαιοσύνη για τις κρατικές προμήθειες, τους διαγωνισμούς ε, και τη διαφθορά στην ανάθεση κάποιων έργων. Χρειάζεται πολιτική βούληση για ε, να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Έχει γίνει πρόοδος βέβαια. Αυτό φαίνεται στη λειτουργία κάποιων εξαρτήτων θεσμών και οργάνων, όπως είναι το ε, θέμα ενός διαμεσολαβητού, του συνήγορου του πολίτη Επίσης γίνονται καλές προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Βελτιώνονται οι σχέσεις με την Κροατία και το Μαυροβούνιο και η Σερβία ε, θα αποτελέσει και θα και μεγάλη πρόκληση για να προχωρήσει και η υπόθεση της Μακεδονίας, λέει ο μιλητής, που περιμένει 6 χρόνια να ανοίξουν τα κεφάλαια. Έχουμε τώρα περισσότερες χώρες ε, με καθεστώς ε, υποψήφιας χώρες. Ελπίζω να παίξει και επικοδομητικό ρόλο το Βελιγράδι για την υπόθεση της Βοσνίας ε, Ερζεγοβίνης. Θα πρέπει να παραμείνει η χώρα ως πολυσυλλεκτικό κράτος, πολυεθνικό, πολυθρησκευτικό και να μην διαλυθεί, να πληρώνει τα κριτήρια και να ενταχθεί κάποια στιγμή ως χώρα η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Χρειάζεται τη βοήθεια της Σερβίας σε αυτό και ελπίζω το συντομότερο να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία, κεφάλαια 23 και 24, δικαιοσύνη, θέματα εσωτερικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή προοπτική να γίνει ορατή για όλους τους πολίτες της Σερβίας. Η μεταρρύθμιση αυτή θα δώσει ελπίδα για καλύτερη ζωή ε, στους πολίτες, ε, οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο για το σύνολο των Δυτικών Βαλκανίων. η Σερβία είναι σε θέση να το επιτύχει όλα αυτά και επιτέλους ε, είναι και προς το συμφέρον των πολιτών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σερβία θα πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας διχάζει και αύριο στην ψηφοφορία ελπίζω αυτό να διαπιστωθεί. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Thank you, President. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κάτσιν, το οποίο είναι εξαιρετική η έκθεση, εξισορροπημένη, πολύ ε, όρημη και εστιάζει την προσοχή του στα σωστά σημεία. Νομίζω ότι σιγά σιγά η Σερβία πλησιάζει το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ε, βέβαια, είναι μακρά η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει και κατά τη γνώμη μου έχουμε ε, την έκθεση η οποία τονίζει το κράτος δικαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τα δε κεφάλαια 23 και 24 είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτή τη διαδικασία βεβαίως. Ε, όπου να θα γίνουν εκλογές, το να πει το αποτέλεσμα βέβαια δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Ε, Ενδεχομένω έχουμε μια τελείως και καινούργια κυβέρνηση η οποία θα αναλάβει τα ενία της χώρας και να δούμε τελικά μέχρι ποιο σημείο το κεκτημένο τη προηγούμενη κυβερνήσεω θα το αναδεχθεί η νέα κυβέρνηση. Κάτι γνώμη μου, θα πρέπει επομένω να πω πάρα πολύ σοβαρά αυτή την έκθεση γιατί τη αξίζει, διότι θα στείλει στη Σερβία ε, τα μηνύματα που πρέπει. Και βεβαίω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή τη Νοτολική Ευρώπη. Η Σερβία είναι πολύ σημαντική ούτως ώστε να πετύχει μια μακρόπνοη σταθερότητα η Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον της χώρας και αυτό θα ωφελήσει επομένω την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κάτσιν για την ισόρροπη και επικοδομητική έκθεση του. Η έκθεση αυτή μας φτάνει σε μια στιγμή αρκετά κρίσιμη. Διότι το Συμβουλίο καλό θα ήταν να ακολουθήσει τη χθεσινή σύσταση και να απονείμει το καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Σερβία λόγω της πρόοδου που έχει επιτελεστεί. Πρόοδος των τελευταίων ετών χάρη και στη συνεργασία της Σερβίας με, το, με διεθνείς φορείς αλλά και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Βεβαίω, η συμφωνία της περασμένης εβδομάδας μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας προκειμένου να υπάρξει μια μορφή περιφερειακής συνεργασίας επί της ουσίας επιτρέπει την ε, συμμετοχή του κοσμοπεδίου σε τοπικά φόρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια έχουμε τεράστιες προσδοκίες για το πώς όλα αυτά θα ολοποιηθούν. Στην ουσία βρέθηκα στο Βελιγράδι μαζί με την αντιπροσωπεία της ομάδας μου όταν υπεγράφει αυτή η συμφωνία Είχαμε οργανώσει μια επίσκεψη εκεί και ήταν σαφές ότι οι αρχές και ο πρόεδρος Τάντζιτς γνωρίζουν τι προσδοκίες υπάρχουν και τι εντυνόμενη ζήτηση εφόσον υπάρξει η απόδοση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία και εφόσον το αποφασίσει αυτό το ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι κάτι που είπε ο πρόεδρος Στάτιτς που είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να το τονίσω. Ότι ο αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος που έχει ξεκινήσει από την κυβέρνησή του είναι προτεραιότητα. Ελπίζουμε και γνωρίζουμε, και εκείνοι γνωρίζουν ότι γνωρίζουμε, ότι θα πρέπει τα κοινά κριτήρια να εκπληρούνται και στην μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και σε όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των μειονοτήτων και όλες τις άλλες πτυχές της λειτουργίας της ίδιας του δημοκρατικού συστήματος και των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου αλλά ακόμη και το πώς λειτουργεί σε συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού η εσωτερική αγορά. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, διότι η απόφαση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Η ερώτηση είναι εάν θα υποστηρίξουμε όσους στη Σερβία είναι υπεύθυνοι για, όλες αυτές τις, για όλα αυτά τα βήματα πρόοδου, προκειμένου να εκπληρώσουν τα κριτήρια της Κοπενχάγης και να στηρίξουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, Διότι πραγματικά πρόκειται για μια χώρα που είναι ευρωπαϊκή δύναμη και ανήκει ξεκάθαρα στην Ευρώπη. Ή εάν θα σφίξουμε το χέρι αυτών που ενώ ισχυρίζονται ότι έχουν ευρωπαϊκό κατάλογο προτεραιοτήτων δεν έχουν κάνει τίποτα. Το αντίθετο. Και πρόσφατα μάλιστα ανησύχησαν διότι η κρίση του ευρώ επηρεάζει και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση τη δική του χώρα. Αυτού δεν θέλουμε να του ενισχύσουμε, γι' αυτό και η απόφασή μα είναι καθοριστική σημασία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το Συμβούλιο θα ακολουθήσει και τι συστάσει του εισηγητή μας για τα θέματα αυτά. Η υπεύθυνη συγγήτριά μα για το θέμα αυτό το μεταξύ δεν μπόρεσε να είναι δυστυχώ σήμερα, γι' αυτό παρουσίασα εγώ την δική τη παρέμβαση λίγο πολύ. Μια από τι παρατηρήσεις της είναι ότι θεωρεί το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σταθερό και συνεπέ στι πολιτικές του τοποθετήσεις. Και να παραμένει πίσω στην του διμερεί ζητήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ω πρόσχημα και ω εμπόδιο για τη διαδικασία ένταξη και στην περίπτωση άλλων χωρών, αλλά ιδίω τη Σερβία. Κοιτάξτε, η κατανομή της εργασίας είναι εξής. Φραντσέσκα Μπράντενερ είναι υπεύθυνη για τη Σερβία. Όμως επειδή έγινε αλλαγή στα θέματα δεν μπόρεσε να παραστεί. Τέλος πάντων, εκ μέρου και των δύο να σας πούμε ότι θεωρούμε πως ε, είναι πάρα πολύ θετικό, ότι πήρε το πράσινο φως η Σερβία, είναι τώρα υποψηφία και επομένως ήρθε η ώρα η Σερβία να κάνει το επόμενο κρίσιμο βήμα στη διαδικασία της προσχώρησης και η επανάληψη των συνομιλιών για το Κόσοβο είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Έχουμε επομένω τέτοια πρόοδο στις σχέσεις ε, των δύο χωρών. Ε, έτσι προλύνεται το έδαφος. Άλλο θετικό είναι ότι τα Γκάλοπ Σερβία ε, λένε ότι τώρα, τώρα που είναι υποψήφια η χώρα θα, θα, θα, ο κόσμος θα γίνει πιο φιλοευρωπαίος. Πιο σημαντικό είναι αυτό μέσα από τις συνομιλίες με την Βελιγραδίου Πρεστίνα και τελικά νομίζω ότι θα, τα ευρωπαϊκά συστήματα θα κατησχίσουν τον εθνικιστικό. Έχει κλείσει το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο μου. Χωρίς μικρόφωνο. Move to that one. Move to that. Oh, yeah. That one works. Right. Okay, yeah. Α, μάλιστα. Α, βρήκαμε ένα μικρόφωνο που να δουλεύει. Έλεγα λοιπόν ότι θεωρώ πως είναι πάρα πολύ θετικό ότι στην Σερβία η προοπτική της ένταξης κάτι ισχύει του, του εθνικισμού. Και αυτό θεωρώ είναι πάρα πολύ θετικό. Και τώρα επομένως θα κάνει αυτό το επόμενο βήμα για την προσχώρηση στη Σερβία θα μπορέσει να δουλέψει περισσότερο για, τους, για τις μεταρρυθμίσεις και λοιπά και ο ανέφερε συγκεκριμένα πού χρειάζεται να γίνει μεταρρύθμιση ε, και ιδίω όσον αφορά τα κεφάλαια 23 και 24 ελπίζουμε ότι εκεί πέρα θα σημειωθεί σύντομα κάποια πρόοδος. Και κάτι θα γίνει σε σχέση με τα σημεία που εμεί έχουμε ζητήσει να δώσουν το βάρο, δικαιοσύνη, ανθρωπινά δικαιώματα, διαφθορά. Επίση, θα πρέπει να συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο στη σχέση με το κρυσφοπέδιο. Έχουν το Σύμβασμα Παριθμών 4 και θα ζητήσουμε χωρίς τη ψηφοφορία εκεί που λέει για το διοικητικό τάδε στην τελευταία φράση. Μιλούμε εδώ για σύνορα, διαχείριση σύνορων. Δεν θέλουμε ότι λογικό να λέμε εδώ πέρα γιατί αυτό το χαρακτηρισμό διοικητικό πρόκειται για σύνορο, σύνορα. Ε, εδώ θέλουμε πάνω στην ψηφορία, ελπίζουμε θα εγκριθεί. Κατά τα άλλα, είπαμε, πάρα πολύ θετική έκθεση και πάρα πολύ θετική, βέβαια, και εξέλιξη τη Σερβία. Ελπίζουμε θα συνεχιστούν τα πράγματα έτσι. Κούκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κάζη τον εισηγητή. Αξιόλογη ε, η έκθεσή του, το σχέδιο έκθεση, αλλά επίση τον ευχαριστούμε και για το πώ συνεργάστηκε με του οικειώδει ηγητέ και με του άλλου συναδέλφου και έτσι θα καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο το οποίο θα μπορούσε να συγκεντρώσει την ευρύτερη συνένεση. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό. Επίσης, να συγχωρούμε τους Σέρβους για τις ε, επιτυχίες τους για το χαιρετισμό της χώρας και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο μπορεί να επικυρώσει όλα αυτά. Έχει τώρα μια αυθεντική ευκαιρία η Σερβία, ώστε να μπορέσει να κάνει αυτό το κρίσιμο βήμα προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση φέτος. Και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί μια έκθεση που θα στηρίζει αυτές τις ε, φιλοδοξίες. Επομένως θα πρέπει να καταστεί υψίστη προτεραιότητα η ένταξη στην ε, Ένωση και αυτό θα είναι θετικό για τη χώρα και για την ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, δεν για τη Σερβία, όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί ακόμα, ακόμα τα πιο δύσκολα που πρέπει να κάνουν του περιμένουν. Επίσης, νομίζω ότι όλα αυτά θα καλυφθούν μέσω των ε, συμβαστικών τροπολογιών και θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτές. Επίση και για τον διάλογο με το Κόσοβο πρέπει να δούμε τι θα γίνει με διαχείριση συνόρων, τι θα πρέπει να γίνει με τι διπλωματεύσεις γιατί ήδη είχαμε κάποιες σχετικές προσθήκες στις συμβαστικές διατάξεις, αυτό είναι πάρα πολύ επίσης ταυτόχρονα. Ε, να δούμε πώς θα υπάρξει κάποιο είδους ουσιαστική συνέχεια κατόπιν αυτών των συμφωνιών και κυρίως ε, να εφαρμοστούν τα όσα συνεφωνήθησαν και από τους ΜΕΝ και από τους ΔΕ για το κρίσιμο παιδί. Επίσης, θεωρούμε πάρα πολύ θετική θέση του Πρόεδρου της χώρας όσον αφορά το δημοψήφισμα για το Κόσοβο. και ελπίζουμε και οι άλλες αρχές της χώρας να υιοθετήσουν παρόμοια στάση όταν έρθει η ώρα των εκλογών για το βόρειο τμήμα του Κωσυφοπεδίου. Να μην γίνουν ε, κινήσεις από πλευρά Σερβίας που θα μας οδηγήσουν σε προβλήματα που το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα. Για την τελευταία φορά που είναι εκλογέ θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια ε, στις φιλοευρωπαϊκές χώρες, τη φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις τη χώρα ώστε να εξασφαλιστεί το ευρωπαϊκό τη μέλλον μέσω των εκλογών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ το λόγο για να πω όσα ήδη υπόθηκαν. Να καλωσορίσω τη συμφωνία μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας με τη βοήθεια της ΥΠΑ της εκπροσώπου και του Επιτρόπου Φίλε, νομίζω ότι είναι μια επικοδομητική προσέγγιση που επιτρέπει στο κοσμοπέδιο να μετέχει στις περιφερειακές συναντήσεις με πολύ συγκεκριμένες διευθετήσεις για το καθεστώς της χώρας. Το συζητώ γιατί προσωπικώς είμαι ευαίσθητος σε ζητήματα καθεστώτος. Αλλά νομίζω ότι εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, τέτοια ζητήματα επιλύονται εύκολα. Και μπορεί κανεί να υπερπηδήσει ακόμη και τα εμπόδια που ακόμη και αν δεν υπερπηδούν μπορεί να παραμεριστούν, να παρακαμφθούν. Εύχομαι λοιπόν η Σερβία να λάβει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, τα τελευταία εμπόδια στο Συμβούλιο να εξαλειφθούν στη Σύνοδο και εύχομαι και καλύτερο μέλλον στις σχέσεις Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ο κ. Πάσκου. Ευχαριστώ. Θα γνωρίζετε ότι η στιγμή αυτή είναι κρίσιμη. Συζητούμε τις προοπτικές μια σημαντικής χώρα της Ευρώπης για το κατά πόσο μπορεί να γίνει να λάβει το καθεστώ υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, ακούσαμε να εκφράζεται η δυσαρέσκεια χθε στο Συμβούλιο. Μάλλον, ακούσαμε να είναι κάποιοι δυσαρεστημένοι, γιατί χθε στο Συμβούλιο υπήρξαν επιφυλάξει ω προ το... αυτή την προοπτική. Και επειδή γνωρίζω τουλάχιστον καλά την περίπτωση μια χώρα που έχει εκφράσει επιφυλάξει, να σα πω ότι η απόφαση αυτή δεν έγινε δημοσίως. Ούτε διαβουλεύσει υπήρξαν και μόνο το μάθαμε μέσα από τα δημοσιεύματα του σερβικού τύπου. Όταν ζητήσαμε διευκρινήσεις, διευκρινήσεις δεν δόθηκαν. Θελήσαμε να καταλάβουμε και τη συλλογιστική της θέσης αυτής, διότι δεν υπήρξε κανένας διάλογος. Θελήσαμε να καταλάβουμε ποια είναι, ποιος είναι ο συλλογισμός εδώ, γιατί δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα αισθήματα των ανθρώπων της χώρας αυτής. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι μένει μετέωρο ένα μεγάλο ερωτηματικό στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που έχει υπάρξει ιδιαίτερα ενεργή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιλύσει το σοβαρό πρόβλημα μεταξύ Σερβίας και Κοσφοπεδίου. Μας φαίνεται λοιπόν κάπως άδικο για τους Σέρβους αυτό, γιατί πάντοτε ήταν μια χώρα φίλη προς το Κωσυφοπαίδιο, προς τη χώρα μάλλον την οποία υπενήχθηκα προηγουμένως. Και μην ξεχνάμε ότι η χώρα εκείνη πριν κάποια χρόνια είχε υποβάλει και εκείνη αίτηση για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως ε, ενδείξεις που αποστέλλονται για το Σέγγεν. Αυτό θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως μια εξήγηση. Αλλά δεν μπορεί κανείς να διορθώνει κάτι στραβό με ένα άλλο στραβό. Ελπίζω λοιπόν, και αυτό ήθελα να εκφράσω εν τέλει, ότι η θέση αυτή θα μεταλλαχθεί και η επιφύλαξη θα αρθεί. Διότι οι μόνοι που μπορεί να επιλύσουν ένα τέτοιο ζήτημα είναι οι ενδιαφερόμενες πλευρές. Εάν ε, πρόκειται να αποσταλεί ένα μήνυμα προς τους Σέρβους, αυτό νομίζω έχει ήδη συμβεί. Έχει ήδη αποσταλεί. Και επίση θα πρέπει να βεβαινόμαστε ότι η παρακολούθηση των υποψήφιων χρόνων για το σεβασμό των δικαιωμάτων και το καθεξής θα διαρκέσει, διαρκέσει, το γνωρίζουμε αυτό και από την ίδια μας την εμπειρία. Ελπίζω λοιπόν, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι οι επιφυλάξεις θα αρθούν και ότι η θέση της συγκεκριμένης χώρας, που δεν θέλω να κατονομάσω, θα μεταλλαχθεί. Ευχαριστώ. Ε, in, in private we can discuss and... ε, μπορώ κατηδίαν να την κατονομάσω κιόλα ημέρο, αλλά όχι εδώ. Ο Λούνατσεκ, Η κυρία Λούνατσεκ, μπορείτε να με βοηθήσετε να τον καταλάβω. Ποια χώρα ήτανε, ας το προσπαθήσω. Ε, μήπως η χώρα του κυρίου Πάσκου, λέω τώρα, εάν αυτό εννοείται πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κατσίν για την έκθεσή του και τις συμβαστικές τροπολογίες. Το έργο του είναι πραγματικά άριστο. Ανέφερε διάφορες σημαντικές πτυχές και επειδή και εγώ είμαι η συγκεντρία υπεύθυνη για την έκθεση του κοσμοπεδίου, θα ήθελα να επικεντρωθώ στα ζητήματα του διαλόγου, το ότι έχει επιτελεστεί πρόοδος και το τι θα πρέπει να κάνει ακόμη η Σερβία στο μέλλον για το ζήτημα αυτό. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για τα αποτελέσματα του διαλόγου την περασμένη Παρασκευή και για τη σύναψη συμφωνίας χθε. μεταξύ Σερβίας και Κοσμοπεδίου. Κανείς δεν θέλησε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα της μελέτης, της μελέτης που έχει γίνει ως τώρα, ότι δηλαδή, της έκθεσης μάλλον που, και των προσμάτων της, ότι ακόμη μένει αρκετή πρόοδος να επιτελεστεί στην ε, Σερβία. Θα πρέπει να γίνει σαφές στη σερβική κυβέρνηση για τις εκλογές ότι οι εκλογές οι τοπικές δεν μπορούν να γίνονται στο βορρά του κοσφοπεδίου. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεν θα πρέπει να οργανώνονται πλέον τέτοιε εκλογέ. Έπειτα, η υλοποίηση τη συμφωνία ε, δεν είναι κάτι το ολοκληρωμένο. Είμαι βέβαια και πεπισμένη ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά τις σερβικές εκλογές. Υπάρχουν ζητήματα όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια που δεν έχουν καλυφθεί. Απομένουν λοιπόν εκκρεμότητε. Επίσης, η συμμετοχή του κοσφοπεδίου για ίδιο λογαριασμό, όπως λέγεται και στη Συμφωνία Διαλόγου. Θα πρέπει να το αποδεχτεί και η Σερβία και οι πέντε που δεν αναγνωρίζουν το καθεστώς της χώρας. Ακόμη και οργανισμοί όπως ο ΑΣΕ είναι περιφερειακοί οργανισμοί. Νομίζω λοιπόν ότι το κοσυφοπαίδιο θα πρέπει να εκπροσωπεί τον εαυτό του στο μέλλον. Υπάρχει λοιπόν κάποια πρόοδος ως τώρα και το να γίνει η Σερβία υποψήφια χώρα θα σημαίνει πολλά για αυτούς, για το λαό της χώρας. Νομίζω ότι το καθεστώς αυτό πρέπει να τη αποδοθεί. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κατά πόσον οι προσπάθειες μεταρρύθμισης και υλοποίηση των κριτηρίων θα είναι ειλικρινής και τίμια στο μέλλον, διότι η ευρωπαϊκή πορεία σημαίνει μια πορεία διαρκούς ε, προσπάθειας και σύγκρισης. Αυτά είχα να πω σε σχέση με το κοσυφοπαίδιο και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για την έκθεσή σου. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου και εμένα μια σύντομη παρατήρηση Νομίζω καλό είναι που λαμβάνεται τώρα η απόφαση να δοθεί καθεστώς υποψήφια χώρα στη Σερβία, διότι θα συνεισφέρει σημαντικά στη σταθεροποίηση της περιοχής και δίνουμε αυτό το θετικό μήνυμα, αλλά θα πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί. Γι' αυτό είχαν επιφυλάξει ορισμένε χώρες ότι και στις συμβιβαστικές τροπολογίες το λέμε, έχει ευθύνη, υποχρέωση η Σερβία να έχει ρόλο και εμφάνιση με τριοπαθή. Και ε, να κοιτάξει ε, τι γίνεται με τις σερβικές μειονότητες που επιτίθενται οι εκπρόσωποι μειονοτήτων που επιτίθενται σε διεθνείς οργανισμούς, σε γραφεία περιφερειακών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε πρόσφατα. Και θα πρέπει ε, να ξέρουμε ότι είναι μια απειλητική αυτή η κατάσταση. Αν δημιουργηθεί εντύπωση ότι η Σερβία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της και δεν δρά υπεύθυνα. Το θέμα δεν είναι η αναγνώριση του κοσφοπεδίου, αλλά κατά πόσο μπορεί να δρά κατευναστικά και να επηρεάζει την κατάσταση η Σερβία. Να μην υπάρξουν ξανά νέε τέτοιε δράσει που μπορεί να είναι απειλή προ τι αποστολέ Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σε τέτοιες περιστάσεις να τους φέρουμε και ενώπιον των ευθυνών τους. Και να το τονίζουμε και αυτό, διότι έχουμε και εμείς ευθύνη για το προσωπικό που εργάζεται στις αποστολές μας και στα γραφεία μας. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, ότι βλέπουμε τα αυτά τα θέματα. Ο κύριος Αγκουράκης παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, εγώ θα είμαι από εκείνους οι οποίοι θα έχουν τη γνώμη ότι η ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδεινώσει πάρα πολύ την κατάσταση των εργαζομένων είτε είναι βιομηχανικοί εργάτες, είτε είναι αγρότες, είτε είναι ε, ε, υπάλληλοι. Το, μιλάω, ε, το λέω αυτό με την εμπειρία της Ελλάδας. ξέρουμε ότι ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται από μια ακόμα μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση, ξέρετε οι προοπτικές είναι για μείωση της ανάπτυξης για αρνητική ανάπτυξη του χρόνου στο 0,3%, ο λαός της Σερβίας πρέπει να σκεφτεί ε, σε τι συμμαχία μπαίνει, σε τι ένωση μπαίνει. Ε, επίσης ε, νομίζω ότι το αντίτιμο που καλείται να πληρώσει ο λαός της Σερβίας είναι πάρα πολύ ψηλός. πλήρωσε μια φορά με τον πόλεμο εναντίον του από τον πληρώνει τώρα στην ουσία με, την, ε, ένα καινούριο βήμα όσον αφορά την απόσχηση του Κωσόβου. Διότι η συμφωνία για την οποία γίνεται λόγος, η πρόσφατη συμφωνία για την ε, συμφωνία της Σερβίας για συμμετοχή του Κωσόβου σε περιφερειακές ε, συναντήσεις και περιφερειακές δομές, δεν αποτελεί τίποτα άλλο από το ότι ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση αυτή και το ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Από εκεί και πέρα το, το κεντρικό ζήτημα που υπάρχει για την ε, ε, χώρα, την ε, γείτονο χώρα, είναι ακριβώς το θέμα της ανάπτυξης. Και αν υπάρχουν αντιδράσεις που αφορούν είτε την παρουσία της K4 είτε της Ulex, αλλά ιδιαίτερα της K4 στο Κόσοβο, αυτή είναι πάρα πολύ απλό να εξηγηθεί. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κόσμος εκεί πέρα αισθάνεται αυτή τις δυνάμεις ως δυνάμεις κατοχής και καλά κάνει και αντιδρά, διότι κανένα λαό δεν αισθάνεται καλά κάτω από ξένη κατοχή και σα φέρνω και το παράδειγμα το πρόσφατο του, του Αφγανιστάν αυτό που γίνεται ε, αυτή την εποχή εκεί πέρα. Κατά συνέπεια, ε, οι Σέρβοι καλό θα κάνουν να μείνουν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αλλιώ θα του κατηγορούν στο μέλλον για ό,τι κακό και ό,τι στραβό θα γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φταίνουν αυτοί, όπω συμβαίνει σήμερα και όπω κύριε Πρόεδρε, δράτουν τη ευκαιρία να καταγγείλω τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος απειλεί τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα εν των εκλογών, ότι όσα δεν συμφωνούν με τις περικοπές και την πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα, ε, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay, thank you very much, Mr. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Κατσίν για την έκθεσή του. Είναι πραγματικά ε, σωστός ο τόνος και η κατεύθυνση νομίζω. Είμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης για την οποία, την οποία δεν πίστευε κανείς, ωστόσο έχει εμφανιστεί. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση και η Σερβία ε, μπορεί να πληρεί ε, τα κριτήρια πλέον και τα πληρεί και της δίνονται ε, τα ειχέγγυα για το καθεστώς ε, της υποψήφιας χώρας. Ελπίζω αυτό να βοηθήσει τις πολιτικές εξελίξεις να σταθεροποιήσει τη χώρα και την περιοχή και θα είναι και προς το συμφέρον ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, ε, Πρόεδρε, σημειώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη θετική τάση στην παρουσίαση και τις αντιδράσεις της έκθεσης του κυρίου Κατσίν. Η πρόοδος της Σερβίας υπήρξε σε κάποια σημεία εντυπωσιακή. Επίσης, θεωρώ και σημειώνω το γεγονός ότι ο κύριος Κατσίν αναφέρει ότι η προηγούμενη έκθεση είναι παροχημένη από πολιτική άποψη και κάποιε τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν και να υποστηριχθούν. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κατσίν. Οι προφορικέ τροπολογίε θα στηριχθούν. Και νομίζω κατά τρόπον ώστε να γίνει πραγματικά πιο επικαιροποιημένη η έκθεση και να, ένα χρήσιμο πολιτικό εργαλείο για την, έκθεση, για την απόφαση που πρόκειται να ληφθεί. Ελπίζω ότι στο Συμβούλιο μεθαύριο θα επιβεβαιωθεί το καθεστώς υποψήφιας χώρας της Σερβίας. Και ελπίζουμε ότι η επιβεβαίωση αυτή, το καθεστώς αυτό, θα ωφελήσει ιδιαίτερος όχι μόνο την Σερβία την ίδια, αλλά την ευρύτερη περιοχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θα θέλαμε να σταθεροποιηθούν επιτέλους τα Δυτικά Βαλκάνια και να ενταχθούν, να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή του ένταξη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρί τη Σερβία. Ακούσαμε κάποιου φόβου να εκφράζονται και από τον εισηγητή και από κάποιου άλλου συναδέλφου ότι κάποια διμερεί ζητήματα θα μπορούσαν να γύρουν νέε ανησυχίε και εμπόδια στην πορεία τη ε, ε, Σερβία προ την Ευρώπη. Όμως νομίζω και ελπίζω ότι η φόβη αυτή ε, δεν είναι βάσιμη. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της χώρας στην οποία κατονόμασε ο κύριος Πάσκου, αλλά βάσει των πιο πρόσφατων ειδήσεων που μόλις το σήμερα το πρωί έλαβα και χθε το βράδυ, νομίζω και προσδοκώ ότι η Ρουμανία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και θα στηρίξει την ευρωπαϊκή μοίρα της Σερβίας εδώ και το είχε κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει και εδώ δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρανόηση. Όμως, να κλείσω λέγοντας ότι για όλους μας αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο μάθημα. Μια χώρα, κράτος μέλος που είναι συνεχώς αντικείμενο άδικης μεταχείρισης, δεν μπορεί διαρκώς να συμπεριφέρεται τόσο λογικά γενναιόδωρα και, και με τον ίδιο τρόπο που έκανε και στο παρελθόν. Βεβαίω και καταλαβαίνω τους φόβους που εκφράστηκαν και ως ένα βαθμό τους συμμερίζομαι. Όμως νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το πρόβλημα αυτό θα ξεπεραστεί το αργότερο μεθαύριο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άρα το συμπέρασμά μου ότι είναι όντως η Ρουμανία, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάουιτ. Και εγώ να εκφράσω το σεβασμό μου για το έργο του κυρίου Κατσίν. Και πραγματικά ήταν εξαιρετική η συνεργασία μεταξύ των διαφορών συνεργατών, υπευθύνων εκπροσώπων. Όπως είπε ο κύριος Κατσίν, στη συζήτηση αυτής της εβδομάδας θα πρέπει να πείσουμε. Δεν είναι απλώς ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα στάδια μιας κλασικής διαδικασίας, όχι. Είναι κρίσιμη συζήτησή μας για την ίδια τη χώρα αυτή και για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν ε, υποστηρίξουμε αυτήν την ε, πορεία τους, θα είμαστε άδικοι και προς τους εαυτού μα και προ τι χώρε αυτέ. Θα πρέπει λοιπόν να περάσει το μήνυμα προ το Συμβούλιο αρκετά ηχηρό και να καταλάβουν ότι θέλουμε το καθεστώ υποψηφίας χώρα για τη Σερβία. Από τις συζητήσεις μα με τον κύριο Κατσίν χθε και με του εκπροσώπου του Συμβουλίου φάνηκε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε βέβαια την πίεση για να οργανωθεί σωστά ο διάλογο μεταξύ Πρίστινα και Βελιγραδίου. Πιστεύουμε ότι πρόοδος μπορεί να επιτελεστεί, αλλά η πίεση θα πρέπει να συνεχίσει να ασκείται. Τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει και ζητώ από τους συναδέλφους να, είναι, να το έχουν αυτό διαρκώς κατά νου, γιατί είμαι και υπεύθυνο εισηγητής ε, για την ε, πρόοδο τη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ανταγωνιστικέ σχέσει των χωρών τη περιοχή ω προ τι μεταρρυθμίσει και το πόσο γρήγορα θα τι ολοκληρώσουν, πώ θα προχωρήσει η ένταξή του. Εμεί ω Επιτροπή και ω Ευρωκοινοβούλιο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στρέψουμε τη μια χώρα κατά τη άλλη. Καλωσορίζω λοιπόν το καθεστώ υποψηφίας χώρα που ελπίζω να αποδοθεί στην Σερβία και σα ζητώ τη βοήθειά σα για να με βοηθήσετε να επηρεάσω και την επιτέλεση πρόοδο στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Ευχαριστώ κύριε Μπρισάτζιτ. My... Όχι. Δεν ήθελα να λέω στον σα. Όμω άκουσα αυτό το οποίο εσεί είπατε και μου γέννησε κάποια ιδέα που θέλω να σα πω. Τώρα καταλήξαμε ότι πρόκειται για τη Ρουμανία βέβαια. Αυτό είναι καλό. Ήθελα να ξεκαθαριστεί. Ναι, ε, πρόκειται για τη Ρουμανία. Και εγώ δε θα ήθελα να ξεκαθαρίζουμε τα εξή δύο. Η Σερβία δεν είναι η χώρα η οποία έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα, ούτε η μόνη χώρα που έχει προβλήματα με τις μειονότητες. Δεν λέω ότι δεν έχει πρόβλημα η Σερβία και ότι δεν επιδέχεται η κατάσταση βελτίωση, αλλά δεν είναι η μόνη χώρα που έχει τέτοιο πρόβλημα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αυτό και για να φρενάρει την πορεία προσχώρησης της Σερβίας στην Ένωση. Τώρα που ξέρουμε ότι πρόκειται περί τη Ρουμανία, επομένω, παρακαλώ συνάδελφοι, όλοι, όλοι, όλοι, κάντε ό,τι μπορείτε. Μιλήστε με του συναδέλφου από τη χώρα αυτή, τη Ρουμανία και ξεκαθαρίστε, εξασφαλίστε ότι οι μειονότητε δεν θα είναι το φρένο στην προσχώρηση. Είναι το θέμα του τι γίνεται σε όλου του άλλους τομείς. Αυτό έτσι να ξεκαθαρίσουμε, Πρόεδρος. Νομίζω ότι θέλετε να κερδίσω σε επόμενε εκλογέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πολύ καλό. Κύριε Κάτσιν, ε, υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Όχι, ο κύριος Κάτσιν. Ε, εάν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα μιλήσω βέβαια εκ μέρου του, αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντα τη λύπη μου που άλλαξε η σειρά εξέταση θεμάτων στην ημερήσια διατάξη και κάποιοι από του συναδέλφου που ενδιαφέρονταν ίσω δεν μπορούσαν να παραβρεθούν. Να αναγνωρίσω ότι όλη η συζήτηση είχε πραγματικά, έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και σε πνεύμα συνένεσης. Συνένεση την οποία καλό θα ήταν να την έχουμε πετύχει πριν επικαιροποιήσουμε το βασικό κείμενο συμπεριλαμβάνοντας τις επιτόπιες θετικές εξελίξεις. Σωστά υπόθηκε ότι οι εκλογές θα διοργανωθούν. Τα πράγματα είναι κάπως απρόβλεπτα, αλλά δεν είναι και η Ρωσία. Η Σερβία Ας ελπίζουμε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και η Σερβία θα λειτουργήσει σε φιλευρωπαϊκό πνεύμα. Βεβαίω δεν ξέρουμε ποιο θα εκπροσωπήσει τη Σερβία στα διάφορα φόρουμ, όμω νομίζω ότι η κρίσιμη καμπή έχει ξεπεραστεί. Το είπα και προηγουμένω, ο διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα ήταν ε, περισσότερο ενδοβελιγραδικό παρά μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Όμω, Νομίζω ότι έστω και αυτή η κίνηση θα πρέπει να είναι κάτι το καλοδεχόμενο από την πλευρά της Σερβίας ε, στο πλαίσιο της, του προκλογικού πυρετού στην ε, Σερβία. Βεβαίως ο διάλογος επικεντρώνεται στο Βελιγράδι, αλλά σίγουρα θα πρέπει να τονωθούν οι προσπάθειες και να συνεχιστούν για το διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Αυτό θα πρέπει διαρκώς να το θυμίζουμε και να το στηρίξουμε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όσα είπε η κυρία Γκόμε. Υπήρξαν κάποιε ανακοινώσει και κάποιε προσδοκίε που εκφράστηκαν από την πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για του πρασίνου και όσε κατά τμήματα ψηφοφορίε έχουν ζητήσει δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα τι δεχτώ. Και για την όλη συζήτηση που έγινε για συγκεκριμένα κράτη, τη Ρουμανία ή άλλε χώρε Ίσως να είναι λιγότερο σημαντικό το πρόβλημα από ό,τι αρχικά πιστεύαμε και νομίζω ότι το τελικό ψηφίσμα θα εγκριθεί. Εδώ καλέσατε του Ρωμάνου συναδέλφου να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Δεν είναι βέβαια στο χέρι του, αλλά στο χέρι τη κυβέρνησή του ή του πρόεδρου Μπασέσκου καλύτερα. Η Μπασέσκου ήταν μαζί μα για κάποια χρόνια. Οπότε νομίζω ότι ο πρόεδρος θα μας δώσει ένα θετικό μήνυμα. και θα γίνει αυτό που όλοι θέλουμε. Τελικώς, ο κύριος Αγκουράκης έκανε μια ομιλία με ιδιαίτερα ιδεολογικό φορτισμένο περιεχόμενο και για την ε, ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά εγώ δεν είμαι υπεύθυνο γι' αυτό. Νομίζουμε ότι η ένταξη της χώρα και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν επικοδομητική για τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί θα έφερναν συνθήκε ασφάλεια σε όλε και θα δημιουργούσαν ένα θετικότερο κλίμα, μια θετικότερη ατμόσφαιρα. Είναι ένα βήμα παραπάνω να περνάει κανεί από το καθεστώ τη γείτονο χώρα στο καθεστώ τη συμμάχου χώρα. Μπορεί να συνεργαστεί έτσι και σε θέματα πιο ευαίσθητα στο μέλλον με τι υπόλοιπε ε, χώρε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την αρμονική μας συνεργασία και να αναφερθώ στο σε όσοι υπόθηκαν για τις προσδοκίες αυτές προς τη χώρα αυτή. Βεβαίως τα προβλήματα μειονοτήτων πάντοτε θα είναι ζωτική σημασία για όλες τις υποψήφιες χώρες ή τις, ε, ε τους, ε, χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση όπως η Σερβία. Όμως σε όλες τις διαπραγματεύσεις υπάρχει περιθώριο όταν περιμένουμε να προστατεύονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Κάποιοι δεν έχουν οργανωθεί ακόμη, κάποιοι μπορεί να οργανωθούν και θέλουμε να ελπίζουμε ότι και εκείνοι θα μπορέσουν να εκλέξουν ε, τους εκπροσώπους τους. Όσες φορές λοιπόν τέτοιες μορφές ε, διοργάνωσης πάρα να δημιουργηθούν θα πρέπει να τις ενισχύουμε και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τις ερβικές αρχές να ξεπεράσουν την κατάσταση που στην αρχή των διαπραγματεύσεων ήταν κάτι που δεν είχε συζητηθεί, αλλά ήταν και κάτι που μπορούσαμε να διαδούμε στον ορίζοντα. Δηλαδή, κάποιες, κάποια κράτη να θέλουν να προστατεύσουν τι μειονότητέ του στο εσωτερικό τη Σερβία. Κύριε Πασκού, σα προειδοποιώ. Από ό,τι θα καταλάβατε από όσα είπα. Even that I have not understood. Ούτε αυτό το κατάλαβα, λέει ο κύριος Μπροκ. Εδώ είναι Βαλκάνια, αγαπητέ μου. Πού να τα καταλάβετε εσείς αυτά τα πράγματα, τα βαλκανικά. Δεν επεξεγέλασε. All very difficult task. Εγώ ένας απλός Βεσφαλός είμαι, τι να καταλάβω από Βαλκάνια. Αλλά ξέρετε τη συνθήκη της Βεσφαλίας ε, και την ειρήνη που ακολούθησε. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε εδώ ε, την πρωινή μας συνεδρίαση. Ραντεβού στις 3 με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, συνεδρίαση, αν δούμε τι γίνεται στην περιοχή. Ραντεβού το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.